Ε, όσον αφορά την εξωτερική πτυχή της ε, Ευρωπαϊκής Ατζέντα για τη Μετανάστευση προς ένα νέο σύμφωνο για την μετανάστευση. Και βεβαίως ξεκινούμε με την Επιτροπή και τον κύριο Τίμερμανς που έχει αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Η Φεντερίκα Μογκερίνη και εγώ είμαστε ευτυχείς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Όπως γνωρίζετε, τους τελευταίους μήνες έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με το ε, Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα των διακινητών που εργάζονται μεταξύ ε, Τουρκίας και Ελλάδας, τις σοβερές απώλειες ζωών στο Αιγαίο Πέλαγος και λόγω των όσων κάναμε το επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των διακινητών έσπασε, ο κόσμος δεν πνίγεται πια στο Αιγαίο και έχει περιοριστεί η ε, κυκλοφορία. Όμως αν δει κανείς στη Νότια Μεσόγειο, ο κόσμος εξακολουθεί να πνίγεται στη θάλασσα. Οι διακινητές βρήκαν ε, άλλη, άλλα περάσματα, οπότε η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο που κάναμε ε, στο Αιγαίο και στη Νότια Μεσόγειο. Να βρούμε λύσεις, βιώσιμες λύσεις. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Η απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε τέτοια κλίμακα και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το σταματήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εμπλακούμε πιο στενά με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, ώστε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της μετανάστευσης σε πρόθεσμα. Αλλά και τώρα άμεσα εμείς και ε, όταν λέω εμείς εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη να μάθουμε από τα διδάγματα του περσινού χρόνου. Σήμερα προτείνουμε μια νέα, ένα νέο πλαίσιο εταιρική σχέση σε συνεργασία με τρίτες χώρες ε, για τη μετανάστευση και ζητάμε από εσά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη καθώ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να στηρίξετε πλήρως αυτή την πρόταση. Το πλαίσιο αυτό βλέπει ξανά πως όλοι οι φορείς, τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι τρίτες χώρες συνεργάζονται ώστε να επιφέρουν την τάξη στις μεταναστευτικές ροές και να προσπαθήσουν για μια σωστή διαχείριση της μετανάστευσης. Θεσπίζεται μια προσέγγιση με προσανατολισμό στα αποτελέσματα ώστε να κινητοποιηθούν όλα τα κράτη-μέλη, τα εργαλεία που έχουν υπόρρητους για αυτό το στόχο προτείνουμε ε, ένα μείγμα θετικών και αρνητικών ε, κινήτρων για να ανταμείψουμε τις τρίτες χώρες που θέλουν να συνεργαστούν αποτελεσματικά μαζί μας και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν συνέπειες για όσους δεν συνεργάζονται. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη χρήση των πολιτικών ανάπτυξης και των εμπορικών πολιτικών ώστε να δημιουργήσουμε μόχλευση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και να είναι έτοιμα να στηρίξουν αυτή την προσέγγιση μέσω των δράσεών τους αλλά και των πόρων τους. Θα δημιουργήσουμε ένα συντονιστικό μηχανισμό ώστε να χειριστούμε πλήρως την συλλογική επιρροή της Ένωσης γιατί μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα. Επιχειρησιακά, βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να σώσουμε ζωές στη Μεσόγειο οι αυξημένε επιστροφέ των όσων δεν έχουν δικαίωμα να μείνουν, να αυξήσουμε μάλλον τι επιστροφέ και να διευκολύνουμε του πρόσφυγε να μείνουν πιο κοντά στι χώρε του και να μην μπαίνουν σε όλη αυτή την επικίνδυνη πορεία. Όσον αφορά τι τακτικές μεταναστευτικέ ροέ, θα πρέπει να ανοίξουμε νόμιμε οδού για μετανάστευση προ την Ευρώπη για όσου το χρειάζονται, ιδιαίτερα με περισσότερη επανεγκατάσταση για του πρόσφυγες. Θα αναπτύξουμε συγκεκριμένε. Ε, συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης, διέλευσης, ανάλογα με τη χώρα, ε, ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τις ε, μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Αυτό θα έχει αποπτά αποτελέσματα για τους πρόσφυγες, για τις χώρες, τις τρίτες που συνεργάζονται και για τι χώρες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προτείνουμε ε, το πρώτα, τις πρώτες συμβάσεις με την Ιορδανία, το Λίβανο, τον Ήγυρα, ε, το Μαλί, τη Συνεγκάλη και την Αιθιοπία. Επίσης, συνεργασία στενή θα έχουμε την Τινησία και τη Λιβύη. Αρχικά θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση της μετανάστευσης επιτόπου στα σύνορα. Αυτό σημαίνει σωστή χρηματοδότηση. Το αφρικανικό καταπίστευμα θα ε, ε, έχει 500 εκατομμύρια από το Αναπτυξιακό Ταμείο αμέσω και ζητάμε από τα κατημέλη να δώσουν άλλο μισό δις. Αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα, να μην περιμένουμε να ε, βουλιάξει άλλο ένα, άλλη μια βάρκα. Θα πρέπει ε, ίσως ε, να κάνουμε περισσότερο από το να κινητοποιήσουμε τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας και να συνδυάσουμε 8 δις αν μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις προσπαθειές μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Αν δούμε τώρα πιο μακροπρόθεσμα τι προκλήσει, πρέπει να κάνουμε περισσότερο ώστε να βελτιώσουμε τι ευκαιρίε τη χώρα προέλευση, ώστε ο κόσμο να μην υποχρεώνεται να φύγει. Γι' αυτό θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα παραδοσιακά μας μοντέλα αναπτυξιακής βοήθεια και να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο ρόλο στου ιδιώτες επενδυτέ. Ενώ οι επενδύσει και η συμφόρηση στις επενδύσει, διαφέρει, μπορούμε, πιστεύω, εκτός Ευρώπης να επαναλάβουμε το επιτυχία του, εσωτερικού, του ε, Ένα νέο δηλαδή ε, επενδυτικό, εξωτερικό επενδυτικό ταμείο που θα έχει στόχο τις, τις επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες αρχίζοντα από την Αφρική και τις γειτονικέ χώρες της Ένωσης. Θα κινητοποιήσουμε 3,1 δις ευρώ που θα αναμοχλεύσουν συνολικές επενδύσεις μέχρι 31 δις και μπορεί να φτάσουμε και τα 62 δις εάν τα κατημέλη ε, συμβάλλουν και αυτά αντίστοιχα. Πιστεύω ότι ε, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και γι' αυτό θα χρειαστεί η δέσμευση όλων των θεσμών, των χωρών και των χωρών εταίρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε είπε και εκπρόσωπος ε, κύριε Μογκερίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να εκφράσω κι εγώ την οδύνη που εκφράσατε χθε για την απώλεια του Τζεν Λούκα Μπορμονάνο. Πάντα είχαμε αντιθέσεις με τον Τζεν Λούκα, έντονες ε, αντιθέσεις, το ξέρετε, όταν και εδώ και στο Ιταλικό Κοινοβούλιο και σήμερα ήταν εδώ παρόν θα βρισκόμαστε σε αντίθετες ε, όχθες, αλλά θέλω μπροστά σε αυτή την τεράστια ονδύνη να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς την οικογένεια, την σύζυγο για τα παιδιά του, τους ε, ανθρώπους τους και την πολιτική του ομάδα. Στα αγγλικά τώρα, για το θέμα που συζητούμε σήμερα. Μαζί με τον Φραντς και τους συναδέλφους στην Επιτροπή έχουμε δύο πολύ σαφή μηνύματα, πολιτικά μηνύματα αφενός και κάποια και πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που ελπίζουμε να τύχουν της πλήρους υποστήριξης του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των υπόλοιπων οργάνων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη μέθοδο. Τους τελευταίους μήνες συζητούσαμε από κοινού τον τρόπο, και αυτός είναι ο τρόπος που θέλει να δουλέψει η Επιτροπή, να προσπαθήσουμε να σε επιτρέψουμε τη σύγκληση των διαφόρων διαστάσεων του έργου μας, προσπαθώντας να δώσουμε ένα στρατηγικό όραμα στις δράσεις μας. Θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο το Φράνς, αλλά και τις υπηρεσίες μας για την εξαιρετική ομαδική δουλειά που πετύχαμε. Το δεύτερο ισχυρό με μήνυμα είναι μια αλλαγή στάσης και παραδείγματος. Πρέπει να περάσουμε από το υφιστάμενο αφήγημα ότι η προσφυγική κρίση και η μεταναστευτική κρίση είναι μια ευρωπαϊκή κρίση στην αναγνωρίση ότι το θέμα δεν είναι θέμα μόνο για την Ευρώπη. Η πλειοψηφία της κίνησης των πληθυσμών γίνεται στο εσωτερικό της Αφρικής και της Ασίας, όχι μόνο προς την Ευρώπη. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μια παγκόσμια προσέγγιση. Ήμουν χθε στη Νέα Υόρκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και συνεργαστήκαμε εν ώψη της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής για τη Μετανάστευση που θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση που προσπαθούμε να παροτρύνουμε. Μια παγκόσμια ευθύνη στην οποία κάθε κράτος, κάθε περιφέρεια, κάθε οργανισμός πρέπει να συμβάλλουν από πλευράς τους. Η Ευρώπη προσπαθεί να συμβάλλει από πλευρά τη, διασώζοντα ζωέ στη θάλασσα. Με την επιχείρηση Σοφία έχουμε σώσει ήδη δεκάδε χιλιάδε ε, ζωέ και οι άλλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο. Όχι μόνο γιατί υπάρχει κόσμο που πεθαίνει στη θάλασσα και πρέπει να σωθεί. Μιλώ και για του χιλιάδε που πεθαίνουν στην Έλληνο πριν, πριν φτάσουν στι ακτέ τη Μεσογείου. Αυτό απαιτεί αλλαγή στην προσέγγιση, αλλαγή στην νοοτροπία που θα μας επιτρέψει να χτίσουμε παγκόσμιες ε, συνεργασίες για να αντιμετωπίσουμε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Τρίτο ισχυρό μήνυμα. Χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στην προσέγγιση μας αφενός στην, στις χώρες της γειτονιάς μας, της Μεσογείου είχαν συμφωνηθεί ήδη συμφωνίες με το Λίβανο το Φεβρουάριο όπου υπάρχει και ένα ισχυρό μήνυμα υλοποίησης. Ένα άλλο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι μια μεγάλη έμφαση στην Αφρική. Η Αφρική για δημογραφικούς, οικολογικούς, κλιματικούς λόγους, λόγω ανισοτήτων θα συνεχίσει να είναι μια σημαντική ήπειρος ότι αφορά τη μετακίνηση των ανθρώπων. Αυτό δεν θα αλλάξει σύντομα Εκτός αν υιοθετήσουμε μια στρατηγική μακροχρόνια προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και τα ζητήματα πολιτικής που είναι στο κέντρο των αιτιών για τους οποίους ο κόσμος εγκαταλείπει τις χώρες τους. Στην ανακοίνωσή μας θέτουμε την σχέση με την Αφρική ή υπόμορφη στρατηγικής εταιρικής σχέσης και βάζουμε και πόρους. Τώρα, δεσμεύσεις. Ο Φραντς ήδη μίλησε για τα κονδύλια. Αύξηση του Trust Fund για την Αφρική, μισό δις ακόμα, συνολικά δηλαδή γίνεται 2,3 εκατομμύρια ευρώ για δράση συναφής με τη μετανάστευση στην Αφρική και θέλω να απευθύνω έκκληση εδώ στα κράτη-μέλη να συμπληρώσουν τις δεσμές αυτές. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και εδώ. Δεύτερον, συγκεκριμένες δεσμεύσεις ανανεωμένες εταιρικέ σχέσεις μέσω των συμφώνων μετανάστευσης και έμφαση σε συγκεκριμένες χώρες. Είπαμε ότι με το Λίβανο ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα τέτοιο σύμφωνο. Πρέπει να το υλοποιήσουμε. Έχουμε εντοπίσει χώρες ε, Νιγηρία, Νίγηρας, Αιθιοπία, Σενεγάλη, Μάλι ως επιπλέον χώρες. Τους τελευταίους 7-8 μήνες ξεκίνησα μια σειρά συζητήσεων με τις χώρες αυτές, κυβερνήσεις, προέδρους, αλλά και κοινωνία των πολιτών και τοπική αυτοδιοίκηση για το τι χρειάζεται στις χώρες εκείνες, σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές των χωρών μερικές φορές, σε χωριά, σε περιφέρειες, όπου, από όπου προέρχονται η πλειοψηφία των ροών λόγω των δύσκολων οικονομικών, κοινωνικών, κλιματικών ή καταστάσεων ή λόγω προβλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικές φορές οι δράσεις μας είναι στοχοθετημένες όταν χρειάζεται και πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση win-win. Να περάσουμε από τη βοήθεια στην επένδυση για την Αφρική, ιδίω ξεκινώντας από τις χώρες εκείνες. Η προσέγγιση του win-win είναι πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο και άρα πρέπει να το διαχειριστούμε από κοινού. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες που είναι χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, η κάθε μία από αυτές πρέπει να έχουν την υποστήριξή μας για να διαχειριστούν καλύτερα τις εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για την διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών με υποδομές και ικανότητα υποστήριξης. Τρίτον, μια μακροχρόνια προσέγγιση, μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Το είπε ο Φραντζ για μια για ένα εξωτερικό επενδυτικό πλάνο που είναι επανάσταση στην αναπτυξιακή συνεργασία της Ένωσης. Το είχαμε συζητήσει με τους Υπουργούς Ανάπτυξης και τους Υπουργούς Εξωτερικών στα δύο τελευταία συμβούλια. Η επένδυση, οι επένδυση στην Αφρική είναι σημαντικό να συνδυάσουμε με έξυπνο τρόπο δημόσιους πόρους της Ευρώπης, ιδιώτες επενδυτές, δεν πρέπει να φοβηθούμε να εμπλέξουμε τους ιδιώτες και διεθνή χρηματοδοτικά ε, ιδρύματα, ιδίω στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καταρχήν. Ακολουθώντα ε, το καλό παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατικών Επενδύσεων, διδασκόμενοι από αυτά που μάθαμε από αυτό και βλέποντα τα επόμενα επενδυτικά προγράμματα που χρειάζονται οι εταίροι μα για υποδομές, βελτίωση των κοινωνικών ε, δαπανών, υποστηρίζοντα την ανάπτυξη στι χώρε αυτέ. Αυτή είναι πιστεύω μια προσέγγιση που είναι ταυτόχρονα και άμεση και στρατηγική. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να συμπληρώσει με συνεκτικό τρόπο τις προτάσεις που είχαν εγκριθεί πέρυσι στην ατζέντα για τη μετανάστευση. Τότε είχαμε μια σειρά μέτρων προς τα έξω. Εμείς επενδύουμε σε αυτό βάση και του τι πετύχαμε στην σύνοδο της Βαλέτα, ενοποιώντας τις ε, προσεγγίσεις μας και εμβαθύνοντας την δουλειά μας και άμεσα και μέσω πρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε με τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Βέμπερ έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Αντιπρόεδροι, η μετανάστευση είναι το σημαντικότερο θέμα αυτής της εποχής και οι συζητήσει που έχουν λάβει η χώρα θα ακολουθηθούν από πολλέ άλλε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν δύο πτυχέ. Από τη μία υπάρχει η εταιρική σχέση, η στήριξη, η βοήθεια. Πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι νεκροί και τα θύματα. Από την άλλη θα πρέπει εμεί να στηρίξουμε τις κινήσεις που έχουν αναλάβει οι Ευρωπαίοι για να σταματήσουν αυτά τα μαζικά κύματα και ροές προσφύγων και μεταναστών. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφές το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Η κατάσταση στα Βαλκάνια ε, δεν είναι πλέον μια έκτακτη κατάσταση ε, ανάγκης. Πρέπει να σταματήσει αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο, στην Μεσόγειο, τα θύματα, οι νεκροί. Ξέρουμε σήμερα όμως ότι η Τουρκία έχει υποδεχθεί πάρα πολλούς πρόσφυγες, εκατομμύρια, και αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να στηρίζουμε, να βοηθούμε την Τουρκία, η οποία υποδέχεται και βοηθάει τους ανθρώπους αυτούς. Την ίδια ώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε επίπεδο ακτοφυλακής προστασίας των συνόρων μας. Και όλα αυτά διότι η απογοήτευση που νιώθουν σήμερα οι άνθρωποι αυτοί όταν ε, θεωρούν ότι μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη είναι μεγάλη. Σήμερα υπάρχει βεβαίως η προσπάθεια για την στήριξη της Αφρικής, το Ταμείο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ξεκάθαρα ότι η δήλωση της Βαλέτα και οι αποφάσεις που λήφθησαν εκεί είναι αυτές τις οποίες θα πρέπει να στηρίξουμε. Βεβαίως και θα πρέπει να έχουμε στρατηγική συνεργασία και εταιρική σχέση με τους γειτονικές μας χώρες. Το μέλλον όμως της Ευρώπης εξαρτάται από την ανάπτυξη της Αφρικής και από το τι θα κάνουμε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σημερινές της προτάσεις. Ευχαριστώ την ε, Φεντερίκα Μογκερίνη, ευχαριστώ τον Φρανς Τίμερμαντ. Πρόκειται για μια πολύ καλή βάση επί της οποίας θα πρέπει να εργαστούμε και να στηρίξουμε τη μελλοντική μας δράση. Επαναλαμβάνω και εγώ ότι ότι θα αυξηθεί εντυπωσιακά ο πληθυσμός της Αφρικής, ότι τα επόμενα χρόνια θα διπλασιαστεί ο πληθυσμός της Αφρικής, είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Και να μην θεωρήσουμε ότι είναι κάτι που μας αφορά περιφερειακά. Πρέπει να επενδύσουμε, πρέπει να επενδύσουμε στην ευημερία της Αφρικής. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα κονδύλια που επενδύονται εκεί. Και αυτό θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε εμείς. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι η Αφρική είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται επικοδομητική συνεργασία γιατί είναι κάτι που έχει άμεση επιπτώσει στην Ευρώπη. Και βεβαίως αυτό το Ταμείο οι προσπάθειες κάθε είδους για εταιρικέ σχέσεις και συνεργασία με τις γειτονικές μας χώρες, αλλά ιδιαίτερα με την Αφρικανική Ήπειρο, γιατί αν παραδείγματος χάρη αρνείται συνεργασία η Αφρική, οι αφρικανικές χώρες, αν δεν δέχονται παραδείγματος χάρη πίσω τους παράνομους μετανάστες, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και εμείς να δούμε πώς θα συνεχίσουμε ή δεν θα συνεχίσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να προσθέσω και μία ιδέα σε αυτήν τη συζήτηση. Η πολιτική μου ομάδα βεβαίως και είναι έτοιμη να δεχτεί τις προτάσεις ε, για την μπλε κάρτα και να είμαστε επικοδομητικοί. Μην ξεχνάτε όμως ότι στην Ευρώπη έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς δουλειά. Στη Νότια Ευρώπη, στις νότιες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν εκατομμύρια νέοι οι οποίοι είναι άνεργοι. Η μπλε κάρτα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι οι συνθήκες αυτών των ανθρώπων θα επιδεινωθούν. Και γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε σαφείς στο μήνυμα που στέλνουμε στους Αφρικανούς που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη η Ευρώπη αυτό μπορεί να το κάνει μόνο από κοινού και μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέμπερ. Όσον αφορά τον επόμενο ομιλητή είναι ο κύριος Πιτέλα. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, συνάδελφοι, ας ε, πούμε την αλήθεια σταθήκαμε μείωπες τα τελευταία χρόνια. Δεν είδαμε ότι ενώπιόν μας υπήρχε μια νέα Ήπειρος με τόσα προβλήματα και τόσες δυνατότητες και κυρίως δεν καταλάβαμε ότι σε αυτή την Ήπειρο με αυτή μάλλον την Ήπειρο, θα μπορούσαμε να έχουμε μοιραστεί αυτές τις προκλήσεις. Αν το σκεφτείτε λίγο, όλες οι μεγάλες προκλήσεις που μας αφορούν, αφορούν και την Αφρική καταπολέμηση τρομοκρατίας. Ε, γίνεται καταπολέμηση τρομοκρατίας χωρίς την Αφρική. Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μπορούμε να την πετύχουμε χωρίς την Αφρική. Διαθρησκευτικός διάλογος. Ανάπτυξη οικονομική, πολιτιστική, ε, ε, πολιτική είναι για μας ετέρωση η Αφρική. Τουλάχιστον τώρα υπάρχει μια καμπή και η καμπή γίνεται χάρη στην Ιταλική κυβέρνηση και χάρη στην Ιταλική Επιτροπή, στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγχωρείτε, χάρη στην Φεντερίκα Μογκερίνη, το Φραντ Τίντερμανς και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάω αμέσως στα συγκεκριμένα. Το, ε, ε, ποια είναι τα προβλήματα. οικονομική πόρη. Κάνατε ό,τι μπορούσατε. 500 εκατομμύρια. Α, αυτό μπορούσατε να κάνετε ρεαλιστικά. Τώρα τα κράτη-μέλη πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δεν μπορούν να λένε και μετά να μην δίνουν τα χρήματα και από πλευρά των κρατών μελών. Και στη συνέχεια έχουμε τον μηχανισμό πολλαπλασιασμού και μόχλευσης ε, επί το οποίο θα πρέπει να επαληθεύσουμε καλά, σωστά. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική ε, Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να είναι μέλος της διαχείρισης της διακυβέρνησης, αλλά πρέπει να αλλάξει και την εντολή της. Δεν μπορεί να χρηματοδοτεί μόνο projects με τριπλό α, γιατί διαφορετικά projects με τριπλό α στην Αφρική δεν, δεν υπάρχουν και γελιοποιούμεθα. Κοροϊδευόμαστε. Τα projects στην Αφρική είναι επικίνδυνα. Άρα τριπλό α δεν έχουνε. Δεύτερο θέμα. Πολιτικής και πολιτιστικής φύσης. Το κόμπακτ αυτό το σύμφωνο, δεν είναι μόνο ε, για την ασφάλεια. Όχι, θέλει να διαχειριστεί καλά τις μεταναστευτικές ροές. Και προσοχή αυτά που λένε ότι οι νέοι Αφρικανοί έρχονται να βουτήξουν τις δουλειές από τους νέους Ευρωπαίους. Μα δεν είναι καν επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό. Ας μιλήσουν αυτοί που τα μελετάνε όλα αυτά. Αυτό το να εξυπηρετούν την ασφάλεια βέβαια, αλλά και το να ε, υπάρξει μια πολιτική, οικονομική και ε, πολιτική και πολιτιστική συνεργασία με την Αφρική. Αν είναι μόνο ένας, μια στρατηγική για να σταματήσουν οι ροές, ε, δεν χρησιμεύει τίποτα. Αν αντιθέτω είναι, όπω είμαι πεπισμένο πω είναι, ένα μέσο ώστε επιτέλου να υπάρξει μια μεγάλη συμμαχία, είναι σπουδαίο εγχείρημα και πρέπει να ε, το ονομάσουμε μια επαναστατική καμπή. Ευχαριστώ, η κυρία Στίβεν, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, πρόεδρε η Επιτροπή έχει ένα <clears throat> master plan για να δώσει χρηματοοικονομική βοήθεια σε χώρες ε, που αλλάζουν ε, πολιτικά στην Αφρική. Το χρειαζόμαστε αυτό όχι μόνο για να χτυπήσουμε την διακίνηση αλλά και την παράνομη μετανάστευση και την επιστροφή αυτών που έρχονται παράνομα. Εμείς ζητούμε λοιπόν οι χώρες ε, της Μεσογείου να συναντηθούν και να κουβεντιάσουν το θέμα αυτό. Γίνεται, ακούσαμε προτάσεις για επιστροφή μεταναστών σε διάφορες χώρες ε, όπως η Τινησία, το Μαρόκο αλλά ταυτόχρονα ε, λέμε να ενσωματώσουμε τους πραγματικούς πρόσφυγες. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοδιοφυλακή θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε με πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ ο κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Να πω καταρχήν στην Επιτροπή ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο με την ε, προσέγγιση τους, με τις συνολικές τους θέσεις ε, που υπέβαλαν σήμερα το πρωί, το νέο σύστημα ασύλου, το, τις νέες προτάσεις για την ακτοφυλακή νέες οικονομικές προτάσεις για την μετανάστευση. Το 1999, αγαπητοί φίλοι, ήμουν παρόν στο Τέμπερε στην Βόρεια Φιλανδία και εκεί πήραμε τις πρώτες αποφάσεις ε, για την πολιτική αστήλου και μετανάστευσης. 17 χρόνια αργότερα, τι βλέπουμε, ότι η κατάσταση που μας απασχολεί σήμερα είναι αυτή που όλοι γνωρίζετε. Όσον αφορά λοιπόν αυτές τις προτάσεις, καταρχήν πρέπει να πω ότι τις θεωρώ καλές. Το θέμα τώρα της επιλογής χωρών για την μετανάστευση. Το θέμα, αν θέλετε, της επικάλυψης της συμφωνίας που υπογράψαμε με την Τουρκία. Ειλικρινά, αγαπητοί Συνάδελφοι, έχω θέμα με αυτό. Έχετε την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Το αποτέλεσμα βέβαια για μας είναι ότι ναι, από αυτήν την οδό λιγότεροι άνθρωποι φτάνουν στην Ευρώπη. Ναι, από άλλες βέβαια οδούς αυξήθηκαν οι αριθμοί. Από την ίδια θάλασσα περνούν, από τη Μεσόγειο. Για τους πρόσφυγες, σίγουρα η λύση αυτή δεν είναι ικανοποιητική. Πάνω από 100.000 πρόσφυγες βρίσκονται εγκλωβισμένοι μεταξύ του Ισλαμικού κράτους και ενός τείχους που χτίζει η Τουρκία και Καταλαβαίνετε ότι ενώ εμείς έχουμε κυρώσει όλες τις ε, συμφωνίες που παρέχουν από τη Σύμβαση της Γενέβης, η κατάσταση είναι δραματική, είναι προβληματική. Δεν είναι λοιπόν λύση η συμφωνία με την Τουρκία για το θέμα αυτό. Και αυτό που μας ζητάτε εδώ να κάνουμε είναι να πολλαπλασιάσουμε τέτοιου είδους συμφωνίες που υπεγράφησαν με την Τουρκία και με άλλες χώρες. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να προσφέρουμε χρήματα για να κρατήσουν στις χώρες τους τους πρόσφυγες. Χρειάζεται πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και των χωρών αυτών. Θα πρέπει από κοινού εμείς με τις χώρες αυτές να δημιουργήσουμε κέντρα υποδοχής στις χώρες αυτές, να τους υποδεχτούμε στην Λιβύη, στην Αίγυπτο, στην Τινησή, στο Λίβανο, στην Ιορδανία, στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και να διαχειριστούμε από κοινού αυτά, αυτούς τους καταβλισμούς, αυτά τα κέντρα υποδοχής και κατόπιν να δούμε ποιοι από αυτούς θα έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως στις χώρες από που έχουν φύγει οι άνθρωποι αυτοί ή στις χώρες τις οποίες βρίσκονται να δημιουργήσουμε δυνατότητες επαγγελματικές και να τους δώσουμε μια ελπίδα να μπορέσουν να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι άλλο. Σε αυτές τις χώρες από τις οποίες περνούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα πρέπει όχι απλώς να τους δώσουμε χρήματα χρήματα εξάλλου που τους είχαμε υποσχεθεί στο παρελθόν που ποτέ δεν τους δώσαμε και σήμερα τους λέμε κρατήστε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και εμείς θα σας δώσουμε τα κονδύλια που σας είχαμε υποσχεθεί. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, χρειάζεται κοινή διαχείριση των συνόρων αλλά και κοινή διαχείριση των κέντρων υποδοχής και των καταβλισμών στις χώρες αυτές. Τέλος, το θέμα της μπλε κάρτας. Ένα θέλω να σας πω. Αυτή η μπλε κάρτα υπάρχει. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι η καλύτερη λύση αυτή θεωρώ ότι θα πρέπει αντίθετα να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει στις Ηνωμένε Πολιτείε. Μία πράσινη κάρτα υπάρχει στις Ηνωμένε Πολιτείε και μία μπλε κάρτα θα πρέπει να δημιουργήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία, ένα σύστημα και όχι 28 διαφορετικά συστήματα και 28 διαφορετικές μπλε κάρτες. Κύριε Σπινέλη, ευχαριστώ. Το Migration Contact αναφέρει πέντε φορές τον όρο δικαιώματα. Εσείς ωστόσο μιλάτε για απελάσεις και καλυμμένες. Λέτε ότι η συμφωνία με την Τουρκία έσωσε ζωές, ζωές αλλά απλώς οι νεκροί πήγαν αλλού. Χιλιάδες πέθαναν το Μάιο στην Μεσόγειο. Λέτε ότι πρέπει να προστατεύετε τους φυγάδες, δίνετε βοήθεια σε 16 χώρες της Αφρικής, αλλά κάθε οικονομική συνεργασία τίθεται υπό την αίρεση του επαναπατρισμού και του ελέγχου των συνόρων των χωρών αυτών. Η βοήθεια που προτείνεται είναι ένα δικτάτ. Ή κρατάτε τους πρόσφυγες σε δικές σας, ε, σε δικές σας προσφυγικές φυλακές ή δεν ε, βοηθάμε. Αυτοί που βιώνουν πολέμους στη Συρία, το Αφγανιστάν, δεν είναι χειρότερη από τις δικτατορίες ε, της Ερυθρέας ε, ή του Σουδάν ε, που δεν πήραν τόσα ωραία δώρα όπως η Τουρκία. Λέτε ότι οι πρόσφυγες πρέπει να γίνουν πιο ανθεκτικοί, αυτάρκεις, να μείνουν σε χώρες προέλευσης ή στις χώρες διέλευσης. Δεν ξέρω αν ξέρετε γιατί μιλάτε όταν ξεδιάντροπα χρησιμοποιείτε ψυχολογικά την αντοχή. Αυτοί που δημιούργησαν κάτι τέτοιο και κατηγορώ καταρχά την Ιταλική κυβέρνηση πιστεύει ότι έχει καθαρά τα χέρια και την καρδιά του. Αυτό έλεγε και η Λέδη Μάκβεθ πριν καταλάβει τι έκανε. Η συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων των διεθνών, των δικαιωμάτων ανθρώπου είναι η είναι, είναι εμφατικά στη συμφωνία με την Τουρκία. Υλοποιείται κύριε, κύριε Τίμερμανς, κυρία Μογκερίνη, πολιτικές που σκέφτηκαν στην Ευρώπη τα πιο ακραία μυαλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάξας. I'm sorry. Uh, my... Οθόνη, Σαρτζεντίνη. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, Κύριε Τίμερμαντς, συνάψαμε μια νέα συμφωνία με την Τουρκία και τώρα μιλάμε για ένα new deal με τις αφρικανικές χώρες όπου προσπαθείτε να αποφύγετε τους πνιγμούς, τους νεκρούς στη θάλασσα και να χειριστείτε τη μετανάστευση. Θα κάνουμε δηλαδή τα ίδια λάθη όπως με τη συμφωνία με την Τουρκία. Δεν λέμε στην Αφρική, βλέπουμε τα προβλήματά μας, βλέπουμε ε, και τα προβλήματά σας και θα δούμε πώς θα σας βοηθήσουμε, πώς θέλετε να σας βοηθήσουμε. Όχι, τα πάντα στηρίζονται περισσότερο στην πρόληψη και όχι στη βοήθεια την πραγματική. Και όταν βλέπουμε τα νούμερα, η Κομισιόν θα πετύχει αυτούς τους στόχους. Έχουν ήδη γίνει μέχρι στιγμής ε, ε, έχουν ήδη γίνει μετρήσεις χιλιάδες νεκροί πέρσι και φέτος. δεν πρόκειται για μετανάστες που πρέπει να προστατευτούν μόνο, αλλά για ολόκληρους πληθυσμούς που πεθαίνουν. Γιατί φεύγουν από την Αφρική οι άνθρωποι. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπάς περιπτώσει, τουλάχιστον είπατε και δύο λόγια για νόμιμη μετανάστευση. Αυτό με κάνει, με χαροποιεί. Ε, ταυτόχρονα όμως θα απειλείται να κόψετε την αναπτυξιακή βοήθεια ενώ είναι εντεταγμένη στην συνθήκη της Λισαβόνας που πρέπει να βοηθήσει τον το κόσμο όμως θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα για να κρατήσετε τον κόσμο εκεί Μα κύριε Τίμερμαν, αν, Τίμερμαν, αν μου το επιτρέπετε, εγώ μιλώ με έναν σοσιαλδημοκράτη, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κανείς δεν μπορεί να ζήσει κλείνοντας τα σύνορα. Και ο κύριος Σίμιτσα, τι, άποψη έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης όταν ε, ε, τα μέλη της Επιτροπής του ΟΣΑ, το μόνο που θέλετε είναι να εμποδίσετε τον κόσμο να έρθει. Ε, οι στόχοι της χιλιετίας δεν έχουν ε, σχέση με όλα αυτά. Η αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είπατε στην εισήγησή σας ε, όσον αφορά τους ε, στόχους σας. Είπατε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίε να μην σεβαστούμε το 0,7% για την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Όμως εδώ χρειαζόμαστε αυτά τα κονδύλια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την Ευρώπη και όχι για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Υπήρξε ένα πρόβλημα στα γερμανικά. Από ό,τι φαίνεται τώρα διορθώθηκε. Next speaker is Mr. Ο κύριος Πάξας είναι ο επόμενος ομιλητής. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να αγοραστεί από κανέναν η ακυρεότητα και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να εξαγοράσει τις χώρες της Δυτικής Αφρικής έτσι ώστε να σταματήσουν οι ροές των ανθρώπων. Αυτό δηλαδή που συνέβη με την ε, Τουρκία, μα είμαστε αφελείς αν νομίζουμε ότι θα είναι αποτελεσματικό αυτό το σύστημα. Τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν, θα δοθούν και τελικά είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που περιμένουμε. Τι να σας πω, είδατε ότι δεν μπορέσαμε να εμποδίσουμε τους τρομοκράτες να έρθουν στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και αλλού και να χτυπήσουν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπα από την αρχή της μεταναστευτικής κρίσης, θεωρώ ότι πρέπει να το επαναλάβω. Όσες συμφωνίες και να συνάψουμε με τις χώρες της Δυτικής Αφρικής, πάνω απ' όλα θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Οι χώρες αυτές Βεβαίως θα πρέπει να ζήσουν με ειρήνη και σταθερότητα, αλλά προϋπόθεση για να πετύχει αυτό το σύστημα είναι να υπάρχει αυστηρός και επαγγελματικός έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε κάθε περίπτωση να σταματήσουμε να στέλνουμε μηνύματα ότι είναι ευπρόσδεκτοι οι άνθρωποι αυτοί, ότι θα τους υποδεχτούμε και ότι θα τους προστατεύσουμε. Οι διακινητές συνεχίζουν λοιπόν ε, το έργο τους και εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να ασφαλίσουμε τα σύνορά μας και να πείσουμε αυτούς που είναι διακινητές να σταματήσουν. Θα ήθελα να σας πω και εγώ ότι άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τους ε, δύο αντιπροέδρους της Επιτροπής. Το ερώτημα δεν είναι εδώ αν θέλουμε ή δεν θέλουμε αυτούς τους ε, μετανάστες. Το θέμα είναι ότι αυτό το φαινόμενο υπάρχει και ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως είδατε, και από τη Λιβύη του Καντάφη, αλλά και από την Τινησία του Μπεναλή, εγκαταλείπουν τις χώρες τους και θέλουν να ζήσουν καλύτερα, με καλύτερες συνθήκες στην Ευρώπη. Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη θα συνεχιστούν και βλέπετε ότι οι περισσότερες προσπάθειες να σταματήσουν δεν το πέτυχαν. Βεβαίως οι πρώτοι που τους προσέλκυσαν ήταν η BMW, η Mercedes και η Audi γιατί είχαν φτηνά εργατικά χέρια, τους ε, προσέλκυσαν λοιπόν στην Ευρώπη και σας παρακαλώ πολύ θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η πολιτική την οποία θέλουμε να στηρίξουμε και να ακολουθήσουμε στην Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη συνεχίζει να είναι μία ανοιχτή ήπειρος για όλους όσους ψάχνουν προστασία και ε, καλύτερες συνθήκες ζωής. Το ίδιο έγινε και το 56 με τους Σούγκρους, αργότερα το 68 με τους Τσέχους και πολύ αργότερα με τους Βόσνιους. Βλέπετε όμως ότι οι μετανάστες σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. Περνάνε μέσα από τρία-τέσσερα ε, διαφορετικά κράτη μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Και αυτό γίνεται βεβαίως με τη βοήθεια των διακινητών. Στην ε, Ευρώπη λοιπόν δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες στις ε, περιοχές αυτές έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην έρχονται όλοι χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζαριανόπουλος έχει το λόγο. Όποιος δεν επισκέφθηκε hot spot, κέντρα κράτησης προσφύγων στα ελληνικά νησιά ή ανοιχτά στρατόπεδα στην υπόλοιπη Ελλάδα, μπορεί να παραπλανηθεί από το ρατσιστικό δηλητήριο της ναζιστικής Χρυσής Αυγής και των Ευρωπαίων συμμάχων της. Ας σκεφτεί ο καθένας πώς θα ήταν αν άφηνε τη χώρα του για να γλιτώσει από τον πόλεμο, την εξαθλίωση και να βρισκόταν φυλακισμένος με κίνδυνο απέλασης γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα δεν τον θεωρεί πρόσφυγα να εγκλωβίζεσαι σε κέντρο κράτησης με τα παιδιά σου σε μια σκηνή στο κρύο τη βροχή και τον αφόρητο ήλιο να είσαι πεινασμένο και να πετάς το φαγητό γιατί δεν κάνει ούτε για τα σκυλιά ενώ εκατομμύρια ξεκοκαλίζονται από ιδιωτικέ εταιρείε σύντηση ή με κυβερνητικέ οργανώσει που χρηματοδοτεί αδρά η ευρωπαϊκή ένωση χωρί καμιά προσφορά του. οι πρόσφυγες λένε δεν ζούμε απλά αναπνέουμε δεν έχουμε κανένα μέλλον η συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας καθιστά την τελευταία ρυθμιστή των προσφυγικών ροών που σήμερα εκτρέπονται προς ιταλία με εκατοντάδες πνιγμένους και μέσα σε ένα παρζάρι μπορεί να επαναληφθούν κάνοντας την κατάσταση αφόρητη. Βάλατε μαζί με την ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα το ατοϊκό λύκο να φυλάει τα θύματα του και να υποδαβλίζει εντάσει στα Βαλκάνια. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα καλεί τον ελληνικό λαό μαζί με του πρόσφυγε να παλέψουν για άμεση μεταφορά του από το κράτο με ευθύνη του κράτου και του ΟΗΕ στι χώρε προορισμού του με εξασφάλιση ανοιχτών αξιοπρεπών ανθρώπινων χώρων φιλοξενίας για όσο διάστημα μείνουν στην ελλάδα με όλες τις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες. Thank you. μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σωστή συζήτηση. Εμείς ως πολιτικοί πρέπει να απομακρυνθούμε από την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση και να, το δούμε, και να δούμε τις ρίζες της μετανάστευσης. Η έμφασή μας θα πρέπει να είναι η πρόληψη των καταστάσεων αυτών. Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά απο, απαιτεί μετρημένη ε, συμπεριφορά, αντιμετώπιση με συμπόνια και ευρωπαϊκή προοπτική. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει έμφαση στη γενιά του αύριο. Αυτό σημαίνει ότι και τα κράτη-μέλη, το ακούσαμε αυτό, πρέπει να συμβάλλουν οικονομικά για να βοηθήσουν τις χώρες να αυξήσουν το, τις δυνατότητές τους. Πρέπει να περάσουμε επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, ένα είδος Marshall Plan που θα επιτρέψει στους ανθρώπους αυτούς να ζήσουν εκεί χωρίς φόβου. Προφανώς χρειαζόμαστε και ε, μέτρα επανεισδοχής και προφανώς οι χώρε αυτές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να δεχθούν πίσω τους πολίτες τους. Αυτό πρέπει να ένα κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Ταυτόχρονα πρέπει να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να ε, ασκήσουμε, να δώσουμε έμφαση και στην ε, υλοποίηση της εφαρμογής του νόμου και στην προστασία εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά. Ο κύριος Φλέκενσταν. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως ε, και εμείς στηρίζουμε αυτήν την ε, πρωτοβουλία. Στα, στο γερμανικό τύπο όμως ε, αύριο το πρωί είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε δηλώσεις όσον αφορά την πρόθεσή μας για το τι θέλουμε να συμβεί στη Δυτική Αφρική. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να επενδύσουμε στο περιβάλλον, ε, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην ανάπτυξη και να εμποδίσουμε τους διακινητές ανθρώπων μέσω συνεργασίας και μέσω προστασίας των συνόρων. Πρέπει να διευκολύνουμε την νόμιμη μετανάστευση εκεί που χρειάζεται στην Ευρώπη και να βοηθήσουμε τις χώρες από τις οποίες έχουν φύγει οι άνθρωποι αυτοί να δεχτούν πίσω αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στην Ευρώπη. Κοιτάξτε παραδείγματος χάρη τι έγινε με άλλες περιοχές. Μόνο με μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη εταιρική σχέση και συνεργασία θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Αλλιώς δεν υπάρχει λύση. Δύο πράγματα με ανησυχούν σε αυτή τη συζήτηση. Το ένα είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Το θίξατε κι εσείς. 1,8 δις εκ των οποίων έχουν δοθεί μόνο 18 εκατομμύρια. Δεν πιστεύω ότι πραγματικά τα κράτη-μέλη θα κάνουν κάτι. Είμαι αισιόδοξο, πιστεύω τις προβλέψεις σας, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει με μεγάλη ταχύτητα να προσχωρήσουν στις εκταμιεύσεις των ποσών που έχουν υποσχεθεί. Η δεύτερη ανησυχία μου είναι με ποιον θέλουμε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα στην κάθε χώρα. Μιλάμε για επενδύσεις για ειρήνη, για σταθερότητα. Χρειάζεται όμως και ρεαλισμός. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι δεν μπορούμε εδώ να εφαρμόσουμε το ίδιο μοντέλο σε όλες τις χώρες. One size doesn't fit all. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσαρμοστούμε και να προσανατολιστούμε με ποιον θέλουμε να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Etheridge. Από τον κύριο δεν τη δέχομαι. Ο κύριος Βαν Όρντεν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ χρειαζόμαστε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση με κάποιες προτεραιότητες που είναι η μείωση του αριθμού των μεταναστών που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα ενισχύει και ενθαρρύνει τη μετανάστευση και σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, να μπορούμε να τους στείλουμε πίσω. Βεβαίως έχουμε υπογράψει τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια και κανένας έλεγχος σε αυτήν την μετανάστευση. Ανησυχώ και εγώ πάρα πολύ με αυτήν την φιλελευθερωποίηση Βλέπουμε πάρα πολλούς ε, από τρίτες χώρες να μπαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξεπερνούν το χρόνο παραμονής που τους έχει επιτραπεί. Χρειάζεται συνεργασία των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών. Κυρία Πρόεδρε, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω συνεισφορά των κρατών μελών προς τον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό για αυτήν τη νέα μεταναστευτική πολιτική. Τα κονδύλια πρέπει να βρεθούν εντός του υπάρχοντος προϋπολογισμού. Υπάρχουν προτεραιότητες οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν, δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις. Από εκεί πρέπει να βρεθούν τα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει καλύτερα να συνεργαστούμε με τις τρίτες χώρες ε, ε, στη γειτονία μας ώστε να διαχειριστούμε τα αίτια της ε, μετανάστευσης, να εξασφαλίσουμε ασφαλή και νόμιμη οδό για την Ευρώπη, αλλά και προστασία των όσων χρειάζονται διεθνή συνεργασία. Συμφωνώ με την Κομισιόν με αυτό, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε και να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές. Είναι σημαντικό ότι τρίτες χώρες ε, είναι αδιέξοδο και η Κομισιόν πρέπει να συνειδητοποιήσει πως η συμφωνία, η δήλωση Ευρώπης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Τουρκίας είναι αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί για να παρακαμφθεί ο δημοκρατικός έλεγχος από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου. Να σας εστιάσουμε αντίθετα στη δημιουργία Ενό αξιοπρεπού συστήματο ασύλου που θα βοηθά τους γείτονές μας αλλά ποτέ να μην αναθέτουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες την ευρωπαϊκή ευθύνη, σε τρίτες χώρες μάλιστα. Διαφορετικά αυτή η Ήπειρο, αυτή η Ένωση θα μείνει θα είναι πάντοτε όμοιρος κάποιου. Ευχαριστώ. Κυρία Βεργιά, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, μα κάνετε πολύ ωραία ομιλία, αλλά δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ε, ο κύριο Τίμερμαν ε, ήταν κάπω πιο ψυχρό. Ο κόσμο αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα τη ανθρωπιστική κρίση ε, σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. 20 εκατομμύρια εκτοπισμένοι το 2015 φεύγουν από καταστροφέ και φυσικέ καταστροφέ. Ένα εκατομμύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η πιο πλούσια οικονομική ζώνη. Από τις ε, χιλιάδες μετακαταστάσεις που είχατε υποσχεθεί, μόνο 1500 έγιναν. Ε, και κάνατε αυτή τη συμφωνία με την Τουρκία που, που, ε, και θέλετε να την κάνετε και για την Αφρική. Θα υποχρεώσετε τις ευρωπαϊκές χώρες να επανεδεχθούν τους μετανάστες, λες και δεν έχουν τεράστια ανθρωπιστική κρίση στην Αφρική. 87% των Αφρικανών μεταναστών ε, κινδυνεύουν. Έχουμε χιλιάδες νεκρούς από πέρυσι. Ε, έχουμε ξεπεράσει τις 10.000 από το 2014 σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΙΑ για, προ... για τους πρόσφυγες. Ε, προσαρμοζόμαστε με κινησμό προς όφελος χωρών όπως η Ερυθρέα και το Σουδάν και βλέπουμε ποιες είναι οι καταστροφές που έχουμε προκαλέσει. Δύο λεπτά η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Κάποιοι συνάδελφοι μίλησαν για αντιμετώπιση της φτώχειας, παραβιάσχημα δικαιωμάτων ανθρώπου, εταιρικές σχέσεις, ωραία είναι αυτά, αλλά αυτό που προτείνει η Επιτροπή είναι άλλο. Να χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο που έχει στη διάθεσή η η Ένωση για την εξωτερική πολιτική μόνο και μόνο για ένα σκοπό, να σταματήσει τους μετανάστες και πρόσφυγες στο δρόμο της στην Ευρώπη. Την αναπτυξιακή πολιτική, τις εμπορικές πολιτικές. Δεν έχουμε κυρώσεις για παραβιάσεις των δικαιωμάτων ανθρώπων στις εμπορικές ε, συμφωνίες, αλλά έχουμε κυρώσεις όταν οι χώρες δεν παίρνουν πίσω πρόσφυγε, άτομα που έφυγαν από τη συγκεκριμένη χώρα. Η Επιτροπή θέλει να δώσει χρήματα και σε χώρε όπω η Ερυθρέα. Εκεί ο κόσμο φεύγει για λόγου εύλογου, βασανιστήρια, ε, δουλεία, παραβιάσει των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν τιμωρεί την Ερυθρέα για να σταματήσουν οι παραβιάσει των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά για να σταματήσει ο κόσμο να φεύγει από εκεί. Τι έχει μείνει από την εξωτερική πολιτική της Ένωσης που στηριζόταν στις αξίες αναφέρατε την παγκόσμια ευθύνη. Πολύ σημαντικό. Όντως. Πού είναι ωστόσο η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών τους δεν μπορεί να γυρίζουμε όλο τον κόσμο και να λέμε στις χώρε διέλευση πάτε περισσότερε πρόσφυγες όταν εμείς η πλουσιότερη ήπειρο στον κόσμο δεν κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Πώς μπορούμε να πούμε στην Τουρκία, την Ιορδανία, άλλε χώρε να δεχθούν περισσότερους πρόσφυγες όταν εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε να, να στεγάσουμε ένα εκατομμύριο. Τα λεφτά δεν είναι αρκετά επανεγκατάσταση. Πώς υποχρεώσετε τα κράτη, κύριε, και κύριε Επίτροπε, να δεχθούν ένα σημαντικό αριθμό προσφύγων, εκατοντάδες χιλιάδες εννοώ τον χρόνο και όχι τις 20.000 ε, ε, που υποσχεθήκαν πέρσι και για τους οποίους μόνο 4.000 υλοποιήθηκε. Το πρόβλημα είναι εσωτερικό της Ένωσης. Δεν χρειάζεται να εξωτερικεύουμε το, την λύση του προβλήματος, αλλά να ζητούμε λύσεις μέσα στην Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Φεράρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η πρόταση της Επιτροπής είναι επεξεργασία εκ νέου του Migration Compact του κυρίου Ρέντσι που περιλάμβανε μια μορφή αμφιλεγόμενης συνεργασίας ε, χω, όχι χωρίς ε, ιστεροβουλίες. Το μοντέλο συμφωνίας με την Τουρκία στηρίχθηκε στην ε, έλλειψη εξωπρέπειας. Πάνω σε αυτό στηριζόμαστε για να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας ε, με τις τρίτες χώρες, δίνοντας εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Διακόπτη. Αν πάτε με τέτοια ταχύτητα δεν σας προλαμβάνουν οι διερμηνείς, κυρία συνάδελφε. Λέω, λίγα λέμε για τη μορφή των δικτατορικών κυβερνήσεων που θα πάρουν τις ενισχύσεις αυτές. Την, ε, λίγα λέμε για την διαφθορά στις χώρες αυτές, την αβεβαιότητα και την αστάθεια κάποιων χωρών όπως η Λιβύη. Δύσκολο μπορούμε να φανταστούμε μορφές συνεργασίας με τέτοιες χώρες. Εν γέν λοιπόν, ναι σε μια αναπτυξιακή συνεργασία για τη διάσωση ζώων, χωρίς υποκρισία όμως μιλάμε για βοήθεια σε μια χώρα, σε μια ήπειρο που από την Ευρώπη το μόνο που γνώρισε ήταν εκμετάλλευση και αποσταθεροποίηση. Ευχαριστώ. Thank you. Next speaker, Mr. Ο Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία Μογκερίνη, θέλει να λύσει ένα συνολικό πρόβλημα. Μα κοιτάξτε, είναι γελίο αυτό. Δεν λύνονται τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο εδώ στην Ευρώπη. Η Τσέσου σήμερα κινήσε με το μήνυμα ότι εμείς ε, οι Ευρωπαίοι πρέπει να εγκαταλείψουμε την ευημερία μας και να υποδεχθούμε μετανάστες από την Αφρία. Κοιτάξτε, χρειάζονται βεβαίως επενδύσεις στην ε, Αφρική. Είναι το ίδιο όμως φαινόμενο και το ίδιο σχέδιο με αυτό του σχεδίου Juncker. Και εκεί δεν δούλεψε και εκεί απέτυχε και τώρα θα αποτύχει. Είναι κάτι που πραγματικά μας γελιοποιεί και που δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα. Βλέπουμε ότι ακόμα και αν επενδυθούν πολλά εκατομμύρια εκεί, η γερμανική κυβέρνηση έχει δεχτεί και έχει υποσχεθεί εκατομμύρια και ε, να υποδεχθεί και να επενδύσει. Μα καταλαβαίνετε ότι με τα 62 εκατομμύρια που αντιστοιχούν αυτή τη στιγμή και τα 93 που έχει υποσχεθεί η Ομοσπονδιακή Γερμανία δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε άλλους μετανάστες. Έχετε μία μπλε κάρτα κύριε Πρέσελ. Ο κύριος Έθριτς. Έχετε 30 δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να... Σας συγχαίρω που έχετε το θάρρος της γνώμης σας και παντάτε στις ερωτήσεις μου. Ε, εσείς θεωρείτε ότι θα γιορτάσουμε το ενέκκληση για παγκόσμια ισότιμη κατά ε, μοιρασιά του πλούτου, όπως ε, υπολογίζεται εδώ. Ε, μήπως καλύτερα είναι να κρατήσουμε τα λεφτά μας στις τσέπες μας και να τα δαπανίσουμε στις χώρες μας, ενώ συνάδελφοι ρίχνουν αλλού τα χρήματα αντί να τα κρατούν για τις χώρες τους. Κύριε Πρέτς. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι βεβαίως στην πράξη ο Φρανς Γιώζεφ Στράους θα σας έλεγε ότι οι ψηφοφόροι, κύριε Βέμπερ, του δικού σας ε, κόμματος και σας μίλησα για το προηγούμενο μήνυμα να εγκαταλείψουμε την ευμερία μας προς την Αφρική, να μεταφέρουμε την ευμερία μας ε, στην Αφρική. Σας εύχομαι πραγματικά καλή τύχη για αυτό που θα συμβεί στις 23 Ιουνίου. Κύριος Βόικτ για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πάντα όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε στην Ευρώπη ε, φτιάχνουμε ένα καινούριο σχέδιο. Ο κύριος Τίμερμανς πέρσι τον Οκτώβριο μας είπε για ένα νέο σχέδιο για να μεταφερθούν 160.000 άτομα. Εν τω μεταξύ βεβαίως μιλάμε για 400 περίπου. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσους που, που έχουν μετεγκατασταθεί. Και μας λέτε τι έχουμε καταφέρει στο Αιγαίο και πρέπει να το κάνουμε και στη Μεσόγειο. Τι έχουμε καταφέρει στο Αιγαίο λοιπόν. Πόσοι από τους 22.000 ε, τους 72.000 ε, με συγχωρείτε έχουν μετεγκατασταθεί μέχρι στιγμής. Υποτίθεται ότι θα είχαν μετεγκατασταθεί. Έχουν ε, μετεγκατασταθεί μόνο λίγες εκατοντάδες. Τι κάνετε για αυτόν που προκάλεσε την κατάσταση. Της ΙΠΑ να πάρουν κανένα πρόσφυγα. Και, κυρία Μογκερίνη, καλή διάσωση στη θάλασσα. Αλλά μετά τι θα κάνουμε. Θα, πρέπει, θα τους ξαναπάμε πίσω σύμφωνα με το αυστραλιανό μοντέλο. Σας ευχαριστώ κύριο Σβέρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ε, έγιναν για να περιορίσουν κάπως την ροή ε, των μεταναστών και τώρα προσπαθούμε να βρούμε μια μεσοπρόθεσμη λύση. Η βοήθεια η οποία δίνεται, ε, η οποία είναι αρκετά υψηλή, έχει στόχο να μπορέσουν οι χώρες αυτές να διαχειριστούν καλύτερα την ροή και να προστατεύσουν καλύτερα τα σύνορά τους. Έχουμε λοιπόν κάποια σημαντικά σημεία και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα κάποιος να υποβάλει έτοιμα στην χώρα του. Χρειαζόμαστε επίσης επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Αυτό θα οδηγήσει στο να παίρνουν λιγότερο τον δρόμο για την Ευρώπη. Πλέον με πολύ περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια από ότι οι Αμερικανοί ή οι Κινέζοι να πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί να δίνουμε στις χώρες που εκπληρώνουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις που ξαναπαίρνουν πίσω τους υπηκόους τους και συνεργάζονται στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Ανεύθυνες κυβερνήσεις που δεν συνεργάζονται δεν πρέπει και να τους ε, δίνουμε και βοήθεια από πάνω ούτε εμπορικές ε, διευκολύνσεις ούτε διευκολύνσεις βίζες. Ο κύριος ε, Σάνι έχει μία μπλε κάρτα για σας. Ναι, έχετε το λόγο. Köszönöm ε, ε, ε, Σας ευχαριστώ. κύριε συνάδελφε, μιλήσατε για την ανάγκη επενδύσεων σε χώρες προέλευσης των μεταναστών. Έχω δύο ερωτήσει. Θεωρείτε ότι το σχέδιο Juncker θα μπορούσε να επεκταθεί σε τέτοια, και σε τέτοια επενδυτικά προγράμματα. Δεύτερο. πιστεύετε ότι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων για τι εξωτερικέ σχέσει και καλύτερη χρηματοδότηση αυτών των χωρών είναι μία λύση. Uh, uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, γεγονός είναι πως υπάρχουν τέτοιες είδες ε, υποτίθεται ότι είναι το σχέδιο Juncker 2 για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι φυσιολογικό ότι χωρίς επενδύσεις από το εξωτερικό και ειδικά ευρωπαϊκές και η Ευρώπη συνεισφέρει περισσότερο στην ε, διεθνή και βοήθεια από την Αμερική ε, δεν θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στις χώρες αυτές και θεωρώ πως ένα τέτοιο ταμείο μακροπρόθεσμα είναι η καλύτερη ιδέα και το σημαντικότερο μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφευχθούν αυτές οι ροές. Ευχαριστώ. Κύριε Παντσέρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η επιτυχία της ευρωπαϊκής δράσης εξαρτάται από μια σειρά συνθήκων. Θα πρέπει να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική που να βασίζεται στην νομιμότητα, την αλληλεγγύη και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης θα πρέπει να έχουμε αξιόπιστους εταίρους. Και το λέω και στο συνάδελφο Βερχόφστατ, ότι για να έχουμε πραγματικές εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να έχουμε λιγότερο φιλελευθερισμό, νέο φιλελευθερισμό στις εμπορικές σχέσεις. Επίσης χρειάζονται πραγματικές ε, χρηματοοικονομικές βάσεις. Αυτό το είδαμε ε, με τη συζήτηση σήμερα χωρίς την παρουσία του Συμβουλίου, δυστυχώς. Καλύτερα να είχαμε προωθήσει τα ευρωμόλογα, αλλά εάν ε, λάβουμε υπόψη τα δικά σας δεδομένα, ας μην έχουμε μία ε, ρήτρα εξασφάλισης. Έχει σημασία να έχουμε τα καταλληλότερα χρηματοοικονομικά μέσα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ο κύριος Μαριάσα, για ένα λεπτό. Είναι δεδομένο ότι στο πρώτο μισό του αιώνα που διανύουμε θα γνωρίσουμε πρωτοφανείς μετακινήσεις πληθυσμών, όχι μόνο λόγω πολεμικών συγκρούσεων η αντιμετώπιση των προσφυγικών αλλά και των μεταναστευτικών ροών πρέπει λοιπόν να αποτελέσει την κύρια κοινή προσπάθεια του οηε αλλά και των κρατών της ευρωπαϊκής ένωσης για τα επόμενα χρόνια. θα πρέπει λοιπόν να χτυπηθούν τα κυκλώματα των διακινητών και να υπάρξει πίεση για την εφαρμογή τόσο τη συμφωνία με την τουρκία η οποία συνεχίζει τους εκβιασμούς όσο και τη συμφωνίας της βαλέτα. αυτό σημαίνει επιτάχυνση των διαδικασιών επαναπροώθησης αλλά και δημιουργία hot spots σε τουρκία λίβανο ιορδανία και σε χώρες της αφρικής για απευθείας επανεγκαταστάσεις προσφύγων στην ευρωπαϊκή ένωση. σε βάθος χρόνου πρέπει να επιβληθεί ρήτρα κατανομής των μεταναστών σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης όπως συμβαίνει και με τους πρόσφυγες. το προσφυγικό και το μεταναστευτικό απαιτούν συνολική προσέγγιση και αυτό σημαίνει πόρους για την αντιμετώπιση της φτώχειας στα αναπτυσσόμενα κράτη καθώς και στήριξη της ανάπτυξης και επενδύσεις στις χώρες της μέσης ανατολής και της αφρικής υπό τον όρο του εκείς σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρίσπεκ για ένα λεπτό ευχαριστώ. Πολλοί είμαστε εμείς που συμμεριζόμαστε την αρχή της συνεργασίας και εταιρικότητας με στοχοθετημένες τρίτες χώρες, κάτι το οποίο είπε και ο κύριος Φερχόφστατ και τόνισε. Σε σχέση τώρα με τις προτεραιότητες που θέσατε για να διασώσουμε ζωές ε, στη Μεσόγειο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 700 άνθρωποι πνίγηκαν πριν από 6-7 μέρες, κάτι το οποίο μας ε, δείχνει ότι το θέμα είναι επίγον. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το εξής. Τη στιγμή που ε, θέλουμε να δημιουργηθεί μία ακτοφυλακή και μία συνοριοφυλακή τάχιστα γιατί ε, δεν θεωρείται ότι η διάσωση θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα της διαφύλαξης των εξωτερικών συνόρων. Είναι ένα από τα αναπόσπαστα στοιχεία δράσης της Frontex μέσα στα πλαίσια και της ακτοφυλακής για τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κυρία Μπιόρκ. Σας ευχαριστώ. Η πρόταση αυτή δεν αφορά ούτε τη συνεργασία ούτε τη μετανάστευση. Απλώς θέλει να τερματίσει τις μεταναστευτικές ροές και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για κάτι τέτοιο. Βλέπουμε πόσο ξενόφοβοι είμαστε και πόσο μας ενδιαφέρει το μέλλον. Φαίνεται ότι καταπατούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα φημώνουμε και μάλιστα συνεχίζουμε να το κάνουμε. Θέλουμε συστηματικά πια να θεσμοθετήσουμε το κλείσιμο των συνόρων και το είδαμε αυτό από τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Φαίνεται ότι οι πολίτες θέλουν μια κοινικά κλειστή Ευρώπη που δεν θα μπορούν να αναπνέουν ενώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα οργανώσουμε μια πιο ανοιχτή Ευρώπη με αλληλεγγύη και να δείξουμε υπευθυνότητα και να δεχτούμε αρκετούς ε, πρόσφυγες. Τερικά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρω ότι η ανταπόκριση μα στην παρούσα ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι σφαιρική. Και πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά υπόψη την κατάσταση στην Αφρική και να τη δώσουμε πολιτική προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά ε, το προτινόμενο σύμφωνο μετανάστευση, θεωρώ ότι παραλείπει δύο εξαιρετικά σημαντικά σημεία. Καταρχήν, δεν αναφέρεται η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πουθενά. Βλέπουμε ενδιαφέρον μόνο ε, να ξεφορτωθούμε τους τωρινούς και μελλοντικού ε, ε, πρόσφυγες και μάλιστα είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε για να τους ξεφορτωθούμε. Δεύτερο θέμα, συναφές και αναπόσπαστα δεμένο με το πρώτο, φαίνεται ότι πιστεύουμε τυφλά και ηθικά και πολιτικά σε όλους τους Αφρικανούς ηγέτες. Ερωτώ λοιπόν, πώς θα εμπιστευτούμε χώρες που αναφέρονται εδώ όπως ε, εμπιστευτήκαμε και την Τουρκία δηλαδή. Θέλουμε να προσπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί χωρίς κάτι τέτοιο, χωρίς ισχυρό δημοκρατικό έλεγχο των διαδικασιών μας και των συμφωνιών μας με τις τρίτες χώρες, θα επαναλάβουμε δυστυχώς όλα τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος. Σας ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Λαβία θέλει να θέσει ερώτηση με την μπλε κάρτα προς τον κύριο Τέρα δεν κάνω λάθος. Ή μήπω όχι. Όχι, κυρία Άτκινσον. Κύριε τερικάβρες, το δέχεστε, ναι. Μιλήσατε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν συμφωνείτε μαζί μου ότι ε, ο κλάδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ουσιαστικά είναι απέναντί μα. Γιατί σε ένα τηλεφωνικό σε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα του BBC, ε, προκάλεσε τον Ερυθρό Σταυρό λέγοντας ότι μετατρέψατε τους οικονομικούς μετανάστες σε πρόσφυγες. Και μάλιστα ήμουνα και στην Ελλάδα πριν από τρεις εβδομάδες και διαπίστωσα ότι τέτοιες ενέργειες γίνεται. Θεωρείτε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων θα πρέπει να τα απαντώνονται σε τέτοιε πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά παντού. Αν κάποιος δεν τα σέβεται, δεν είναι δικό μου φταίξιμο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριος Χούκε, με 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, επειδή έχω δει τις, ε, τις ακτές του Σέγγεν μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα μάνα εξ ουρανού για τους μετανάστες οι οποίοι ε, πηδούν φράκτες και μεταβαίνουν όπου θέλουν. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει τα χρήματα των Βρετανών φορολογουμένων να πάνε σε αυτή την πολιτική. Αν θέλετε να σταματήσετε με τους θανάτους στη ε, Μεσόγειο, τότε θα πρέπει να στέλνουμε πίσω τους μετανάστες. Εμείς έχουμε τη δική μας ε, εισρωή μεταναστών στην Νότια Αγγλία και προσπαθεί αυτό να το ε, αναχαιτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα συζητηθεί στην πρώτη Ολομέλεια μετά το δημοψήφισμα. Γιατί το κάνουν αυτό. Το ξέρουν διότι ξέρουν ότι οι Βρετανοί δεν θα δεχτούν κάτι τέτοιο δηλαδή να εισραίουν ε, μετανάστες με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα ψηφίσουμε στο δημοψήφισμα. Δείτε τι θέλει η Ευρώπη. Θέλει χρηματοδότηση 50 δις. Αυτό είναι ένα άλλος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ψηφίσουμε να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια μπλε κάρτα Κύριε Χούκεμ, έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Μπόγκοβιτς. Τη δέχεστε? Κύριε Μπόγκοβιτς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, 23 και μετά τις 23 Ιουνίου θα υπάρχει οπωσδήποτε μεταναστευτική πίεση. Πιστεύετε σοβαρά ότι μετά τις 23 ε, Ιουνίου θα έχει απαλλαγή από το πρόβλημα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν ε, δεν είστε μέσα θεωρείτε ότι το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του χωρίς να συνεισφέρουν οι Βρετανοί. Κύριε Χούκομ. 23. 23 Ιουνίου. Ελπίζω όταν φύγουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το λύσει από μόνη της. Εμείς είμαστε νησιωτική χώρα, θα κανονίσουμε τα δικά μας σύνορα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φοντάνα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ύπατη εκπρόσωπο για τα θετικά της λόγια. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Βεβαίως υπάρχουν οι μεταναστευτικές ροές και πολλές φορές ε, κερδίζουν οι διακινητές, οι εγκληματίες και στη συνέχεια μετατρέπονται σε τρομοκράτες που εντάσσονται σε ευρωπαϊκές τρομοκρατικές οργανώσεις. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε αυτές τις ροές. Υπάρχει όμως και ένα το δικαίωμα. Ένας άνθρωπος θα πρέπει να μπορεί να ζήσει στη χώρα που γεννήθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε γιατί οι αφρικανικές χώρες εφαρμόσουν πολιτικές ώστε να μην παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στο έδαφος τους και μπορούν να γίνουν συμμαχίες με χώρες όπως η Τουρκία όπου δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό επιφέρει μία και στις δικές μας πολιτικές. Ο κύριος Συναδεινός. Συζητάμε για ένα σχέδιο αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης Αναρωτιέμαι όμω τι απέγιναν τα παλιά. Πέτυχαν ή απέτυχαν. Χρειάζονται επικαιροποίηση ή έχουν καταντήσει παλιόχαρτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο να αναλάβει την ευθύνη και να πει με θάρρο και περισσή αλήθεια το απέτυχε. Να ψελίσει ένα μέα κούλπα. Ω τώρα αποτύχατε εκτρά. Το αποδεικνύουν οι φράχτε στα σύνορα των Βαλκανικών χωρών και η χρήση του άρθρου 25 τη συνθήκη Σέγγεν από τα κράτη-μέλη. Τώρα προωθείται νέο σχέδιο επανεισδοχή με τρίτε χώρε, ενώ το περίφημο σχέδιο επανεισδοχή με την Τουρκία ουδέποτε εφαρμόστηκε προωθείται αναθεώρηση τη μπλε κάρτα για υψηλά κατηρτισμένου λαθρομετανάστε όταν η ανεργία των νέων επιστημόνων διαρκώ αυξάνεται. μιλάτε για ένταξη και απορρόφηση των λαθρομεταναστών όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι προέρχονται από χώρε με νοοτροπία και θρησκευτικέ πεπιθήσει έξω από κάθε έννοια κράτου δικαίου και ειρηνική συνύπαρξη. επιτέλου α αναλάβει κάποιο την ευθύνη αποτυχία. πλέον οι αποτυχημένε πολιτικέ σα βάφονται με το αίμα αθώων ανθρώπων στο παρίσι τι βρυξέλλες την κοπεγχάγη και το αιγαίο πέλαγο πλέον μετρώνται με στατιστικά αυτοκτονιών με ξεριζωμούς νέων ανθρώπων από τις πατρίδες τους με αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και ροπής προς ψυχοτρόπες ουσίες. τέλος θέλω να επιστρέψω στο αιμοσταγές κουκουέ και τον ευρωβουλευτή του τα στα τύπου σχόλια για τη χρυσή αυγή. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εδώ και πολύ καιρό, πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούμε μια πραγματική ένταξη της μετανάστευσης σε εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πραγματική διπλωματία για τη μετανάστευση. Και έχουμε σήμερα την ενοιολογική τουλάχιστον σύλληψη. Η πρόκληση είναι να τη συγκεκριμενοποιήσουμε, να τη δώσουμε σάρκα και οστά. Θα ήθελα να επισημάνω τρία στοιχεία. Πρώτον, μια ευρυθής ανάλυση της χρηματοδότησης είναι απαραίτητη Αφενός των βέλτιστων πρακτικών ε, των χωρών που έχουμε επιλέξει ως κατά θα πρέπει ε, να αξιοποιηθεί και και επιπλέον να δούμε ε, πώ θα χρησιμοποιήσουμε το ΦΕΤ και του χρηματοδοτικού μα μηχανισμού και να μειώσουμε τον ρυθμό των προτεραιοτήτων για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεύτερον, σίγουρα η Αφρική είναι μια ήπειρο κλειδί. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να, ενισχύσουμε τη στήριξη του ελέγχου των συνόρων μεταξύ των Αφρικανικών χωρών και μια διαφρικανική διαχείριση τη μετανάστευσης. Σε ό,τι αφορά του, τα αίτια τη μετανάστευση θα πρέπει οπωσδήποτε ε, με την ε, αναπτυξιακή συνεργασία να πετύχουμε αποτελέσματα θα πρέπει να βρούμε μια προσέγγιση και κίνητρα που θα έχουν κάποια λειτουργικότητα, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εμπορικά ίσω και οικονομικά κίνητρα ε, για να έχουμε μια μόχλευση και ε, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στι υπόλοιπε χώρε που δεν είναι χώρε προτεραιότητα, έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ποιο είναι ο ρόλο των περιφερειακών αφρικανικών οργανώσεων. Επίσης, ε, για το σχέδιο δράσης της Βαλέτας, τι μέτρα προτάθηκαν για να αξιοποιηθεί το δυναμικό ε, της Αφρικανικής Διασποράς ε, στην Ευρώπη και επίσης ε, πώς θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών της Υποσαχάρη Αφρικής και των νότιων χωρών της Μεσογείου και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γκερέρο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Με την υιοθέτηση του μεταναστευτικού πακέτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη γνώμη, υιοθέτησε σωστή προσέγγιση και εστιάστηκε στο σωστό σημείο. Θέλει μια σφαιρική, στρατηγική προσέγγιση, καλύπτοντα τις διάφορες πτυχές της ε, πραγματικότητας μετανάστευσης, που στηρίζεται σε συμφωνίες σύνδεσης ε, με τις ε, χώρες προέλευσης, ε, διέλευσης και προορισμού των ε, μεταναστών και μάλιστα έχει και μέσο και μακροπρόθεσμη προοπτική. 60 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν, είναι εκτοπισμένοι λόγω εμπόλεμων σειράξεων. Είναι λοιπόν προφανές ότι ένας παγκόσμιος εταίρος στην πρόληψη και διευθέτηση των κρίσεων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταπολέμηση της, επανα... της μετανάστευσης γιατί Υπάρχουν άλλα 60 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί λόγω της πείνας και των ανθρωπιστικών κρίσεων. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε επενδύσεις για να θέσουμε ένα τέρμα στη φτώχεια στις περιοχές και χώρες αυτές. Τέλο, ω εισηγητή για την ανθρωπιστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να τονίσω ότι η, όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να δράζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο και στι αρχέ τη ανθρωπιστική δράση. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Κέλμελ. Θα ήθελα να πω ε, προς το εξ του ECR και του κομματός μας να πω πως θεωρούμε πως τα σημερινά μέτρα είναι σωστά. Και βεβαίω θα πρέπει η βοήθεια να πηγαίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στι αιστείε τη κρίση, αλλά και τα συνοδευτικά μέτρα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και τα συνοδευτικά μέτρα είναι σαφώ εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί πέρα έχει αποτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε ενιαία αντιμετώπιση όσον αφορά την διασφάλιση των εξωτερικών μα συνόρων. Δεν έχουμε ενιαία εφαρμογή του δικαίου, κάθε χώρα κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν ακόμα χώρες που λένε ότι εμείς ε, μπορούμε να πάρουμε ανθρώπους ε, απεριόριστα και το κάνουν αυτό. Υπάρχουν άλλοι που έχουν βάλει ε, ποσοστώσεις και άλλοι κάνουν απελάσεις. Και βεβαίως το πώς θα διασφαλιστούν έτσι τα εξωτερικά σύνορα είναι ένα ένιγμα Πρέπει λοιπόν ε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τα του οίκου μας ε, και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε για βοήθεια στην Αφρική. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μλίναρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω το ότι η Κομισιόν δίνει οικονομικά κίνητρα για το θέμα αυτό. Η συμφωνία με την ε, Τουρκία όμω δεν μπορεί να αποτελεί υπόδειγμα. Και ελπίζω να μην περάσουν και αυστριακές προτάσει που μιλάνε για αυστριακό μοντέλο, δηλαδή να πηγαίνουμε τις βάρκες στα διεθνή ύδατα, να ε, έχουμε έγκλειστους ε, ανθρώπους ε, με περιορισμένα ή καθόλου ανθρώπινα δικαιώματα. Πέρα από το εάν κατά πόσον παραβιάζουν αυτά το διεθνές δίκαιο δεν γίνονται και πρακτικά γιατί ποιος Ευρωπαίος ναύτης ε, πολεμικού ναυτικού θα σταματήσει με ποιο πλοίο, ποια βάρκα πριν φτάσει σε κάποιο νησί. Κοιτάξτε, έχουμε κάποιους ε, στόχους, αλλά θεωρώ πως ε, θα πρέπει τουλάχιστον η Αυστρία και οι άλλες χώρες να εφαρμόσουν τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χρυσόγωνος για ένα λεπτό η ευρωπαϊκή επιτροπή κάνει λόγο για ένα σύμφωνο για τη μετανάστευση με κεντρικές ιδέες τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ένωσης και την καταπολέμηση του δουλεμπορίου σε συνεργασία με αφρικανικά και ασιατικά κράτη κατά το πρότυπο της πρόσφατης συμφωνίας με την τουρκία. όλα αυτά όμως αποτελούν απλώς τρόπους προσωρινής διαχείρισης και δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του ζητήματος. οι έντονες μεταναστευτικές ροές οφείλονται αφενός στις απάνθρωπες οικονομικές πολιτικές λιτότητας και στην ανυπαρξία δημογραφικής πολιτικής στο εσωτερικό της ένωσης με αποτέλεσμα η ευρώπη να υποφέρει από δραματική υπογεννητικότητα και αφετέρου στη φτώχεια και τους πολέμους στον ευρύτερο γεωγραφικό μας περίγυρο. χρειαζόμαστε ένα άλλο μείγμα πολιτικής στο εσωτερικό προκειμένου να υποστηρίζεται περισσότερο η ανατροφή παιδιών και η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους και στο εξωτερικό ώστε να επικρατήσει ειρήνη στη μέση ανατολή και τη βόρεια αφρική και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων εκεί. αν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή πολιτικής το πρόβλημα θα επιδεινωθεί περαιτέρω. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σκοτ Κάτω για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δέχομαι τις ανησυχίες που αναφέρθηκαν για τις επιπτώσεις των μεταναστευτικών ροών. Δυστυχώς αυτό επέδρασε αρνητικά στην ε, προεκλογική εκστρατεία για το Βρετανικό δημοψήφισμα. Εμείς ελέγχουμε τα σύνορα μας, γι' αυτό δεν θα θα πρέπει να υποστηρίξουμε το να μπορέσει να μπει η Μαρίν Λεπέν στα δικά μας σύνορα για να μιλήσει ε, στα πλαίσια του δημοψηφίσματος. Επίσης, θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε μαζί τους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, καταστροφικές μας πολιτικές στη Μέση Ανατολή. Ως προς την ελεύθερη ε, μετακίνηση έχει μεγάλη επίπτωση το όλο θέμα στα νοικοκυριά γιατί πρέπει να μπορέσουν να βγουν από τα σύνορά μας και να ε, ζήσουν και να συνταξιοδοτηθούν εκτός Μεγάλης Βρετανίας. One minute. Κύριε Άτκινσον, για ένα λεπτό. Μιλάμε για ένα αφρικανικό καταπίστευμα, δηλαδή να ε, φύγουν τόσα χρήματα και να τα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Μόνο πέρσι δώσαμε 2,5 ε, δις στερλίνες στους Αφρικανούς, δηλαδή οι φορολογούμενοι χρηματοδοτούν και τις ΜΚΟ που εργάζονται κατά της ε, ε, βούλησης των Ευρωπαίων. Ήμουνα με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Μιλήσαμε για άνοιγμα των συνόρων, αλλά και οι ΜΚΟ σοκαρίστηκαν από αυτές τις δηλώσεις γιατί τα δις αυτά δεν θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν τη στιγμή που η βιομηχανία ανθρωπίνων δικαιωμάτων εργάζεται υπέρ των ε, μεταναστών. Θα πρέπει να απορρίψουμε τις ε, προτάσεις σας, να απορρίψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ψηφίσουμε Brexit στις 23 Ιουνίου. Κυρία Άτκινσον, υπάρχει ε, μία μπλε κάρτα από τον κύριο Ζακόφσκι. Την δέχεστε, ο κύριο Ζακόφσκι. Ευχαριστώ. Συμφωνείτε με την άποψη κάποιων ε, που είναι υπέρ ε, του να παραμείνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε ότι όσοι θέλουν Brexit δεν γνωρίζουν τα γεγονότα. Είπατε ότι στην Λίμπε είμαστε υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Πότε πατήσατε τελευταία φορά στην Επιτροπή. Πού ακούσατε αυτά τα πράγματα. Μάτκινσον. Κυρία Άτκινσον. Ήμουν πριν από 15 μέρες εκπροσωπώντας την ομάδα μου στην Λίμπε και συζητήσαμε το θέμα μετά την διάσκεψη των Προέδρων και ζήτησα να μην μπει ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μας αγνόησε η Επιτροπή, ο Τίμωθη Κέρκοπ αρνήθηκε να συζητηθεί η πρόταση της ομάδας μας. Και πριν από τρεις εβδομάδες όταν ήμουν στα στρατόπεδα των προσφύγων, ο κύριος Νίντερ Μιλέρος Σοσιαλιστής είπε ότι έχουμε ανοιχτά σύνορα εμείς ε, Υπάρχουν τρεις ομάδες εδώ μέσα που ήταν σε αυτήν την ε, συνάντηση και είπαν ότι δεν μπορείτε να τα λέτε αυτά, είναι επικίνδυνα. Και οι ΜΚΟ το ίδιο είπαν. Ρωτήστε τους σοσιαλιστές συναδέλφους σας. Το είπαν αυτό και στέλνουν το λάθος μήνυμα στην Αφρική και όλα τα άλλα εκατομμύρια που θέλουν να έρθουν στις χώρες μας, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντέξουμε. Ευχαριστώ κύριο Σκόρβιν Μίκη, Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα, το πρόβλημα δεν έγκυται στην ισροή των προσφύγων, αλλά είναι κατάλληλοι αυτοί οι μετανάστες που έρχονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ε, αυτό που θέλουν είναι περισσότερο επιδόματα οι μετανάστες που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ε, κάποιος ε, πολιτικός μίλησε για τις ε, αφρικανικές ορδές που σειραίων στην στην Ευρώπη και μάλιστα μίλησε πολύ αρνητικά για αυτές τις αφρικανικές ορδές. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτή η πολιτική. Ε, να σταματήσουμε να τους δίνουμε επιδόματα και να τους αναγκάσουμε να εργάζονται. Και μια και ε, με το παράδειγμα θα πρέπει να διδάσκουμε, θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να κόψουμε τα δικά μας επιδόματα πρώτα. Γιατί ο σοσιαλισμός ε, είναι ε, ένα καθεστώς που ε, ουσιαστικά ε, έχει πολύ αρνητικό τρόπο εφαρμογής και νομίζω ότι όλοι εδώ στην αίθουσα θα πρέπει να το διαπιστώσουν. Κύριε Μίκε, θα πρέπει να μας σέβεστε και να μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες, ε, ακατάλληλη ορολογία και εκφράσεις που δεν συνάδουν με το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπλε κάρτα κύριε Μίκε. Τη δέχεστε. Ένας α, Κογκολέζος διπλωμάτης. Κύριε Κόρβιν Μίκε, ερωτώ, τι στοιχεία χρησιμοποιείτε όταν μιλάτε με τέτοιο τρόπο. Έχετε κάποια στοιχεία, πού στηρίζεστε. Ξέρετε ε, Άλλε περιοχέ του κόσμου πώ έχουν κερδίσει με την εκμετάλλευση τη Αφρικανική Επίρου ε, αιώνε επί αιώνων. Θέλω στοιχεία. Όχι απλά λόγια. Ο κύριο Κόρβιν Μίκε. Δεν κατάλαβα καλά τη σχέση έχει ε, τι, τι έγινε, πώς, ε, τι στόχο έχει αυτή η εκμετάλλευση Αφρική. Εγώ μίλησα για το Κονγκό ε, το Παγού ξέρει τη, στη μετανάστευση από την Αφρική προς την Ευρώπη. Ξέρω ότι από τη στιγμή που δίνουμε επιδόματα ενεργείας, ε, ουσιαστικά παξιώνουμε τον κόσμο. Θα πρέπει να καταργήσουμε τα επιδόματα, να στείλουμε τον κόσμο να δουλεύει και όχι να κάθεται και να παίρνει επιδόματα. Ο κύριος για λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε δεν είναι πάντα ευχάριστο να βλέπουμε σε τι βαθμό σουρεαλισμού έχουν φτάσει οι συζητήσεις εδώ μέσα. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με την δήλωση ότι κρίνοντας από τον αριθμό των αναφορών στον καημένο Βρετανό φορολογούμενο από Βρετανούς συναδέλφους που δεν έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής καμία ευρωπαϊκή επιδότηση ε, θα πρέπει να θέλουμε να φύγουν οι άνθρωποι ε, για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους. Ε, Μπα και εξαλαφρώσουν λίγο οι Βρετανοί φορολογούμενοι. Ε, επί της ουσίας τώρα, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω τα εξή. Θα ήθελα να σας πιστέψω, ε, κυρία και κύριε Αντιπρόεδρε, αλλά δεν ξέρω. Δεν, δεν αρκούν αυτά τα πράγματα. Ε, ίσως μια συμφωνία με κάποιες χώρες να αρκούν αυτά. Αλλά για να αναπτυχθεί η Αφρική ή να πάει η δυναμική της Αφρικής σε μια διαφορετική κατεύθυνση, πολύ αμφιβάλλω. Τα 500 εκατομμύρια που υποτίθεται ότι θα πήγαιναν από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο είναι λιγότερα από όσο θα επενδύσουν οι Κινέζοι σε μια σιδηροδρομική γραμμή από τη Μομπάσα στην Κεντρική Αφρική. Αυτό δείχνει ακριβώς ε, τη διαφορά μεταξύ των προθέσεών μας και των όσων είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε όταν πρέπει να κάνουμε τα λόγια μας πράξη. Ε, θα ήθελα να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε μια Αφρικανική αναγέννηση. Αλλά με αυτά τα κονδύλια φοβάμαι ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ευχαριστώ η πρόσφατη τραγωδία στην Κρήτη και στις ακτές της Λιβύης δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση κατεπίγουσας ανάγκης. Όταν έκλεισε ο Βαλκανικός δρόμος, ο μόνος τρόπος πρόσβασης είναι η Μεσόγειος. Οι σημερινές προτάσεις αφορούν μια νέα προσέγγιση στο μεταναστευτικό και νέα συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών προέλευσης και διέλευσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχουν έργα υποδομής που προβάλλονται για τις χώρες αυτές και να βοηθήσουμε και μέσω ΕΙΕΔ. Η Ιταλία ζητά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μεταναστευτικές ροές δεν θα σταματήσουν στο εγγύς μέλλον και πιστεύω ότι χρειάζεται η συμμετοχή όλων γιατί πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι μεμονωμένων κρατών. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ähm, Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπατή εκπρόσωπε. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή επιστρέφει σε γνωστές μεθόδους που χρησιμοποίησε σε προηγούμενες κρίσεις από το Μαρόκο προς την Ισπανία, από τη Λιβύη προς την Ιταλία πριν από μια δεκαετία, εδώ και μια δεκαετία. Πώς να κρατήσει τους μετανάστες εκτός των συνόρων της δηλαδή. Η κυρία Μογκαρίνη μίλησε για αλλαγή του αφηγήματο και ότι ε, η μεταναστευτική κρίση δεν είναι πλέον ευρωπαϊκό αλλά παγκόσμιο πρόβλημα. Σωστό. Ε, σωστό επίσης όμως είναι ότι αντί για βοήθεια στην Βόρεια Αφρική καλό θα ήταν να κάνουμε επενδύσεις. Άλλαξε όμως και το δικό μας αφήγημα για τη μετανάστευση. Ακούσαμε πρόσφατα ότι όλοι οι μετανάστες έχουν μια θέση στην Ευρώπη και ότι θα τροφοδοτήσουν την ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Φοβάμαι όμως μήπως προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους ανέργους στην οικονομία μας που ήδη μαστίζεται από την ανεργία. Και δεν θα πρέπει με το άσυλο να φέρνουμε σε αντιπαράθεση τα κράτη-μέλη. Και μην ξεχνάτε ότι τα εγκληματικά αυτά κυκλώματα δεν θα εγκαταλείψουν ε, το, την προσοδοφόρα απασχόληση της λαθροδιακίνησης. Θα πρέπει περισσότερες επενδύσεις να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε ολιστικά τη μεταναστευτική κρίση και ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο κόσμος όλος έχει δράσει επαρκώς έτσι ώστε οι πρόσφυγες να βρουν έναν ασφαλή λιμένα οι Σύριοι, οι Ορδανοί χρειάζονται να μπορούν να, πολλά ε, μέσα και θα πρέπει τα παιδιά τους να μπορούν να πάνε σε σχολείο. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη βοήθεια στους πρόσφυγες και στα παιδιά τους. δεν μπορεί να δράσουν μόνο τα Ηνωμένα Έθνη. Μόνο έτσι θα απαλληλθεί η κατάσταση στη Μεσόγειο. Διαφορετικά, καμία συμφωνία με την Τουρκία δεν θα βοηθήσει. Οι απελπισμένοι άνθρωποι θα βρουν άλλες οδούς. Αγαπητοί συνάδελφοι, τη στιγμή που μιλάμε για μια νέα μεταναστευτική συμφωνία, η κατάσταση αντί να καλυτερεύει, χειροτερεύει. Καθημερινά αθώοι άνθρωποι, μεταξύ αυτών πολλά παιδιά και βρέφη, καταδικάζονται σε θάνατο μονάχα την τελευταία εβδομάδα του Μαου 900 άνθρωποι πρόσφυγες ξεψύχησαν στη Μεσόγειο. Η κατάσταση είναι ντροπή και απαράδεκτη. Δεν γίνεται η επίσημη πολιτική της Ένωσης να συνεχίζει να καταστρατηγεί τις διακηρυγμένε αρχές της για αλληλεγγύη, να κλείνει τα σύνορα, να προωθεί τις απελάσεις, να υπογράφει ντροπιαστικέ συμφωνίες με την Τουρκία για τους πρόσφυγες. Η κατάσταση είναι τραγική. Ακόμα και οι άνθρωποι που σώζονται από τα πολύ νεκρά ναυάγια βρίσκονται αντιμέτωποι με άθλιες συνθήκες διαβίωσης και με τα hot spots να μετατρέπονται σήμερα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. για να σταματήσει το έγκλημα πρέπει να πάψουν οι κούφιες υποσχέσεις και να ληφθούν άμεσα μέτρα να δημιουργηθεί άμεσα ένα κοινό και δίκαιο σύστημα ασύλου στηριγμένο στην έμπρακτη αλληλεγγύη και την ισότιμη κατανομή βαρό. να δημιουργηθούν νόμιμοι και ασφαλείς οδοί καθώς και ένα μόνιμο δεσμευτικό και δίκαιο σύστημα μετεγκατάστασης των προσφύγων εξίσου σημαντικό είναι να γίνουν ανθρώπινοι και αξιοπρεπείς χώροι φιλοξενίας των προσφύγων τόσο στην ένωση όσο και στις τρίτες χώρες. ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Άνεμανς. Αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπουμε πως ε, οι έχοντες ε, την εξουσία μιλάνε τώρα για ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης το οποίο είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από σύμφωνο. Βλέπουμε πως υπάρχει περαιτέρω επέκταση αυτής της, ε, αυτού του εκβιασμού όπως είδαμε και στην ε, συμφωνία με την Τουρκία και γενικώ παραλλαγές στο ίδιο θέμα. Περισσότερα κονδύλια, περισσότερα λεφτά των φορολογουμένων. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απογοητευτεί. Πρέπει να παραδεχτούμε την αποτυχία της Σέγγεν, την αποτυχία της πολιτικής ανοιχτών συνόρων. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση, χρειαζόμαστε λιγότερη επιτέλους. 1,5 λεπτό, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρωτοφανής αυτή μεταναστευτική κρίση των τελευταίων χρόνων ε, μας έχει πείσει ότι κανένα κράτος μέλος από μόνο του δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Χρειαζόμαστε καλύτερα συντονισμένες κοινέ ευρωπαϊκές απαντήσεις και πιο αποτελεσματική συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Του λεχθέντω θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή ενώ θα πρέπει να ακολουθήσει τις ακόλουθες ε, προτάσεις για να ελαφρύνει την μεταναστευτική κρίση. Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ οικονομικών μεταναστών και προσφύγων. Ε, όσοι αναζητούν καλύτερη ζωή θα πρέπει να ακολουθήσουν τις νόμιμες ε, διάβλους. Βέβαια, κανένα κρατος δεν έχει ένα νομικό πλαίσιο ώστε να αποκρούσει την παράτυπη μετανάστευση δεν θα πρέπει να περιμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει στους παράτυπους μετανάστες την ίδια στήριξη με αυτή που δίνουμε σε πρόσφυγες που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Επίσης, ε, θα πρέπει να ε, ε, επαναπατρίσουμε τους παράτυπους μετανάστες όσους δεν έχουν δικαίωμα να τύχουν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνάψουμε συμφωνίες επανεισδοχής με τις ε, χώρες προέλευσης. Επίσης θα πρέπει να επανεξετάσουμε την ιδέα της ε, συγκρότησης ε, hot spot κέντρων καταγραφής και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελαφρύνοντας την πίεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο σε δικαιούνται η διεθνή προστασία να μπορούν να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από τη στιγμή που έχουν λάβει άσυλο με βάση το ενωσιακό δίκαιο. Η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης χρειάζεται νέα μέτρα και νέα προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας θα είναι απαραίτητο στοιχείο της κοινωτικής δράσης. Καλωσορίζω αυτή την ανακοίνωση. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν προτεραιότητα μέσα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, αλλά υπάρχουν και άλλες ευάλωτες χώρες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έχουμε ε, δώσει 18 εκατομμύρια στο 1,2 δις αυτού του καταπιστεύματος για την Αφρική. Μιλάμε λοιπόν για αναπτυξιακή βοήθεια και επειδή υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, οι κίνδυνοι είναι και ε, μεγαλύτεροι. Αυτά τα ομόλογα δεν θα ήταν χρηματοοικονομικά, αλλά ομόλογα αλληλεγγύης. Γι' αυτό και η Ιταλική πρόταση δεν είναι και πολύ καλή πιστεύω ότι μιλάμε για μία πρόταση και των Ηνωμένων Εθνών μέσα στα πλαίσια του COP21 σε σχέση με ένα ε, φόρο ε, συναλλαγών. Νομίζω όμως ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, δεν μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσεις με ανθρώπινες ζωές, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτό ακριβώς έκανε. Μίλησε για ένα καθεστώς θεωρήσεων που απελευθερώνεται εάν ε, γίνονται δεκτοί άνθρωποι. Το 86% ε, των προσφύγων βρίσκονται στο Νότο και δεν μεταβαίνουν προς την Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε πώς διακινδυνεύουν και να λάβουμε υπόψη και από πού προήλθαν. Εάν μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Αυτή η πρώτη ανακοίνωση δείχνει ότι η πολιτική της ΕΙΕΔ είναι πολύ καλή οικονομικά αλλά όχι πολιτικά θεωρώ ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο διπλωματικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς. Όχι να το κάνουμε μόνο, όχι να το λέμε, αλλά να το κάνουμε. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι είναι δέσμευση της ΥΠΑ της εκπροσώπου και μαζί με τον πρόεδρο Τίμερμανς θα τύχουν τις υποστήριξής μας. Κόρβιν Μίκε έχει ζητήσει το λόγο επί διαδικαστικού θέματος. Παρακαλώ κύριε Κόρβιν Μίκε. Ποιο είναι το διαδικαστικό θέμα που θέλετε να θέσετε. Δεν θέλω να απαντήσω σε κάποιον που έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις προηγουμένως. Ζήτησε το λόγο επί διαδικαστικού. Πείτε μας ποιο είναι το διαδικαστικό θέμα κύριε Κόρβιν Μίκη. in my speech there was used word in word shit. It was not in my it was not not not. Ακούστηκε ε, η λέξη ε, shit στα γαλλικά, περιτόματα. Εγώ μίλησα για καταβόθρες, σάμπο. Αψάω μετά στα γερμανικά. Σκάμ. Όχι shit. Δεν μίλησα εγώ για περιτόματα. δεν φταίω εγώ για τη διερμηνία. Εγώ χρησιμοποίησα την λέξη καταβόθρα ανθρώπινη. Ακούσαμε την δύσοσμη ερμηνεία όσων είπατε. Προχωρούμε στους επόμενους ομιλητές. Ο κύριος Σούλικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Οι πολιτικές ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ αδύναμες για να προστατεύσουν την Ευρώπη. Προτιμούν να πληρώνουν άλλες χώρες για να ξεφορτωθούμε τους μετανάστες. Αυτό είναι και υποκριτικό και επικίνδυνο γιατί μετά εξαρτώμεθα από αυτές τις χώρες. Και εντωμεταξύ βεβαίω ε, την ε, ροή την μείωσε αισθητά το κλείσιμο των ε, συνόρων της υπογνωμού και όχι συμφωνία με την Τουρκία. Έτσι και η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να φυλάξει τα σύνορά της, αλλιώς θα το κάνει η Αυστρία στο στενό του Μπρένερ. Είναι ψευδέστηση να νομίζουμε ότι κάποιος μηχανισμός κατανομής ή κάποιες πληρωμές είναι η λύση. Ναι, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αλλά να τους βοηθήσουμε εκεί. Η πλειοψηφία των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατά της μαζικής μετανάστευσης. Εάν οι σημερινές πολιτικές ελίτ δεν το αντιληφθούν και δεν τα καταφέρουν, οι άνθρωποι θα επιλέξουν εξτρεμιστές. Όχι γιατί ε, αυτό θέλουν, αλλά γιατί θα έχουν αποτύχει και έχουν αποτύχει οι πολιτικές ελίτ. Ευχαριστώ. Μία μπλε κάρτα, κύριε Σούλικα, από τον κύριο Κώστα. Τη δέχεστε? Have a blue card. Παρακαλώ. Κυρία Κώστα. Θα ήθελα ε, όταν λέ, να μου πείτε, όταν λέτε ότι πρέπει να κλείσει τα σύνορα Ιταλία τι σημαίνει αυτό να ξαναρίξουμε στη θάλασσα αυτούς που προέρχονται από τη θάλασσα και από τόπους που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές, γυναίκες, μικρά παιδιά. Πώς να κλείσουμε τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα. Τους ξαναρίξουμε στη θάλασσα. Sie müssen sie nicht wieder zurück ins Meer werfen, auch nicht erschießen. Είπα, ούτε να τους πυροβολήσετε, ούτε να τους πετάξετε στη θάλασσα. Πηγαίνετε τους από εκεί που ξεκίνησαν. Εκεί επιστρέψτε τους. Εκεί πέρα πρέπει να φτιάξει κάποια στρατόπεδα υποδοχής η Ευρώπη, όπως υπάρχουν στη Λιβύη, στην Τουρκία. Όπως υπάρχουν στην Τουρκία πρέπει να υπάρξουν και, στο... και στη Λιβύη. Αυτή είναι η λύση, κατανομή στην ε, Ευρώπη και μετά να τους στέλνουμε πίσω πακέτο. Δεν γίνεται έτσι. Για ένα λεπτό ο κύριος Τέλιτσκα. Στην ουσία η συμφωνία με την Τουρκία ε, άλλαξε τα δεδομένα με τους διακινητές. Βλέπουμε ότι πρόκειται για πιο επικίνδυνο δρόμο και μπορεί να είναι θανατηφόρος. Γι' αυτό το πακέτο σας είναι πολύ θετικό. Έχουμε διαφωνίες, αλλά αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Υπάρχει ε, αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των επενδύσεων, της χρηματοδότησης και με τις μεταναστευτικές ροές, όχι με τις ε, διόδους ροών. Νομίζω ότι το θέμα της Τουρκίας θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, αλλά δεν είναι επαρκές σε αυτό το πλαίσιο αν δεν υπάρχει μία σωστή πολιτική επαναπρόφησης. Θα πρέπει να υπάρξει μία εξισορρόπηση έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειαζόμαστε για μία ευρωπαϊκή λύση και η πόλωση που έχουμε σε άλλα ζητήματα θα ανασυρθεί. Η επίγουσα ανάγκη υπάρχει. Ακούμε αυτά που μας λέει συνέχεια ο κύριος Ρέντσι, κυρία Μογκερίνη. Μας είπατε ότι είμαστε ρατσιστές, ξενόφοβοι. Εσείς στην ουσία δεν κάνατε τίποτα. Μιλάτε αλλά δεν κάνετε τίποτα. Στρουθοκαμιλίζετε. Είπατε ότι οι μετανάστες είναι πηγή ε, πλούτου. Ντροπή σας γιατί είσαστε κοινωνοί αυτής της κατάστασης. Ο κύριος Ρέντσι μιλάει για ένα ε, φλινάφημα όπως ήταν και η πολιτική Γιούνκερ. Κάθε μέρα χιλιάδες παράνομοι εισραίουν στην Ιταλία. Ας μην λέμε ψέματα, ας πρέπει, θα πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα και να, υπερασπιστούμε, και να τα υπερασπιστούμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Ακούγοντας μερικούς ομιλητές, έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν ε, πρόσφυγες ε, εμποδίζουν και τα μέτρα για να μην έρθουν περισσότεροι. Και πραγματικά, κύριε Σούλη, και εσείς εκφράζετε αυτή την υποκρισία. Και τι η συμφωνία με την ε, Τουρκία σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι σταματάμε τους διακινητές και βοηθάμε τους ανθρώπους στην Τουρκία και αρχίζει να λειτουργεί. Πρέπει να το πούμε. Δεν ε, πώς θα γινόταν δηλαδή να τους επιστρέψουμε τους ανθρώπους αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία και διαπιστώνουμε επίσης πως ήρθαν τώρα αυτές οι προτάσεις για να εφαρμοστεί κάτι ανάλογο στην ε, Αφρική όπου είναι πιο περίπλοκη κατάσταση γιατί το πρόβλημα είναι πρόβλημα ανάπτυξης και προσπαθούμε ακριβώς να βοηθήσουμε και να υπάρχουν και ανθρώπινες συνθήκες τουλάχιστον στα στρατόπεδα προσφύγων ε, και βεβαίως να κινηθούμε κατά των διακινητών ε, στην Βόρεια Αφρική. Είναι λογικά σημεία αυτά αφετηρίας. Οι προτάσεις που λέτε εσείς, δηλαδή όταν είναι οι άνθρωποι στη θάλασσα να τους ε, σώσουμε και μετά να δούμε ή να τους επιστρέψουμε στην ε, ακτή. Δεν ξέρω εάν μπορούν να γίνουν. Νομίζω πως είναι ε, η μόνη λογική πρόταση αυτή την οποία βλέπουμε. προκαλέσατε ένα κύμα ενδιαφέροντος για μπλε κάρτα αλλά θα δώσω μόνο μία μπλε κάρτα ως δικαίωμα στον πρώτο κατά σειρά, τον κύριο Κριστέα. Δέχεστε αυτή την μπλε κάρτα. Οι κύριοι Σούλη και Τέλιτσκα σήκωσαν μετά το χέρι τους και έχουν ήδη μιλήσει, άρα προηγείται ο κύριος Κριστέα. Τη δέχεστε. Κύριε Κριστέα, έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Αναφερθήκατε στις χώρες που δεν θέλουν να δεχτούν μετανάστες πώς δέχεστε την θέση του Προέδρου Ιωάννη της Ρουμανίας σε σχέση με το θέμα αυτό της μη αποδοχής. Κοιτάξτε, δεν μίλησα για χώρες, μίλησα για συναδέλφους εδώ μέσα που είναι και κατά των προσφύγων και κατά των μέτρων για να μην έρθουν περισσότεροι πρόσφυγες. Δεύτερον, θεωρώ πως θα έχουμε ούτως ή άλλως λιγότερους πρόσφυγες με αυτά τα μέτρα και ε, θα γίνει πιο εύκολα και μια κατανομή. Κατόπιν, ε, προς τον κύριο Σούλικ, μόνο να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της χώρας, να ε, τελειώσουμε τους πολέμους, να υπάρξει ανάπτυξη, αυτό είναι ο αποφασιστικός παράγον που θα εμποδίσει τους ανθρώπους να βγαίνουν στη θάλασσα. Τώρα το σειρματόπλεγμα στο Μπρένερ ή στα ελληνομακεδονικά σύνορα τι να σου πω, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες του πολιτισμού. Εγώ δεν θέλω να γίνουν στρατόπεδα προσφύγων. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαδάκης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η επιτυχία του νέου συμφώνου για την μετεγκατάσταση δεν έγκυται στη θέσπιση νέων μέτρων για αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης αλλά στην πιστή εφαρμογή του χωρίς παρεκκλήσεις. αλλιώς θα εκτεθούμε και πάλι ως ευρωπαίοι όπως με την εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης όπου υπερτέρησαν οι εθνικοί εγωισμοί. αλληλεγγύη ίση κατανομή βάρους προσήλωση στι αρχέ και αξίε τη ευρωπαϊκή ένωση σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έμφαση στι νόμιμε διόδου μετανάστευση, συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτων χωρών προέλευση και διέλευση, επαρκή και βιώσιμη χρηματοδοτική βάση. αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να διέπουν το νέο σύμφωνο. πρέπει να υπάρχει κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων η οποία θα εξασφαλίζει ασφάλεια καταπολεμώντα παράλληλα εγκληματικέ δραστηριότητε δραστηριότητες. ωστόσο διαχείριση συνόρων δεν συνεπάγεται κλείσιμο συνόρων. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αντιπροέδρους της Επιτροπής για την πρόταση που μας παρουσίασαν σήμερα που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να επανεκκινήσουμε μία διαδικασία επενδύσεων για τις χώρες προέλευσης ε, των προσφύγων για να παραμείνουν εκεί. Αλλά εκεί να υπάρχουν συνθήκες ανάπτυξης για να αναχαιτιστεί η πορεία τους προς την Ευρώπη. Ξέρουμε βεβαίως ότι μέσα σε 30 χρόνια αυτές οι ροές θα γίνουν ολοένα και μεγαλύτερες. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε σταθερές σχέσεις με αυτές τις χώρες. Τα 500 εκατομμύρια δεν επαρκούν, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς μίλησε για μία πρόσμιξη κινήτρων και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα αρνητικά στοιχεία για αυτές τις χώρες της Ευρώπης που δεν συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία και δεν θέλουν να ανταποκριθούν. Όλες είμαστε ευρωπαϊκές χώρες και δεν σημαίνει ότι αυτές που βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα θα πρέπει να καταβάλουν και ολόκληρη την προσπάθεια. Θα πρέπει να υπάρχουν και αρνητικά κίνητρα για αυτούς που δεν συνεργάζονται έτσι ώστε να επιτύχει αυτό το εγχείρημα. Κύριε Λαβία, έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Φρουντζουλίκ. Τη δέχεστε? Κύριε Φρουντζουλίκ, παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε, εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης, της κοινωνικής και των εμφυλίων πολέμων σε μερικές χώρες στην Αφρική, η Ευρώπη θα δεχτεί ολοέτερα και διονγκούμενες ροές, ιδιαίτερα από την Αφρική. Δεν νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει μία μακροχρόνια στρατηγική για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Γιατί δεν πρόκειται για έμπρακτα μέτρα ή πρακτική υφής μέτρα. Χρειαζόμαστε μία μακροχρόνια στρατηγική. η μπλε κάρτα δεν είναι ομιλία Κύριε Λαβία, έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η στρατηγική αυτή δεν είναι βραχυχρόνια, γιατί μιλάμε για επενδύσεις σε αφρικανικές χώρες που δεν θα αποδώσουν βραχυχρόνια. Θα πρέπει να μιλάμε για ένα πακέτο δισεκατομμυρίων το οποίο είναι μακρόχρονο, μακροχρόνιο, μακρόπνο. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε βράχη χρόνια τι πρέπει να κάνουμε πρώτα. Για ένα λεπτό η κυρία Ροντρίγκες. Ε- Ευχαριστώ. Ε, αξιότιμη Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η επιλογή μας είναι σαφής. Είτε θα μείνουμε μια παλιά ήπειρο στην αμυντική θέση, σε άμυνα, είτε θα ε, ξεκινήσουμε μια εταιρική σχέση για το μέλλον με τις γειτονικές χώρες για να στηρίξουμε την ανάπτυξή τους, για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τη μετανάστευση και να στηρίξουμε και τους πρόσφυγες. Το δίλημα είναι σαφές και η επιλογή μεταξύ των δύο. Βέβαια αυτό προϋποθέτει σημαντικές ενέργειες, ε, σημαντικές ενέργειες ε, και κυρίως τις επενδύσεις. Επενδύσεις σημαίνουν και θέσεις απασχόλησης και πολλές νέες θέσεις απασχόλησης μπορούν να δημιουργηθούν και για τους νέους της Ευρώπης αλλά και για τους νέους ε, στις γειτονικέ χώρες. Πιστεύω ότι αυτό το επιχείρημα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία που θα, θα δημιουργηθούν την αυτή πρωτοβουλία. Έτσι θα πείσετε τα κράτη-μέλη να αφιερώσουν και δικού του πόρου στην πρωτοβουλία, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερε συνεισφορέ από τα κράτη-μέλη. Επίση, ε, μέχρι στιγμή οι νέοι το έχουν καταλάβει πολύ καλά αυτό στην Ευρώπη και συμμερίζονται αυτό το όραμα. Έχουν και οι ίδιοι αναλάβει πολλέ πρωτοβουλίε προ αυτή την κατεύθυνση και με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σα αναγγείλω ότι πολύ σύντομα οργανώσει νεολαία θα καταθέσουν συγκεκριμένε προτάσει που θα έχουν ακριβώ αυτή την ίδια κατεύθυνση. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Τέλιτσκα. Αν και ο κύριο Τέλιτσκα μίλησε πριν 10 λεπτά. Κύριε Τέλιτσκα, λέω να μην σα δώσω την μπλε κάρτα, γιατί έχουμε ήδη βγει εκτό χρόνου και μιλήσατε πριν 10 λεπτά. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Πάμε, περνάμε τώρα στον κύριο Ρανζέλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω και είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως ως προς το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται τους διαρθρωτικούς παράγοντες και λόγους. Έχουμε εδώ δύο, δύο μέτωπα. Το άμεσο μέτωπο που είναι ε, το μέτωπο της διάσωσης ανθρώπινων ζώων και θα πρέπει να μην φυστούμε προσπαθειών και μέσων για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, γιατί χάνουμε πολλές ζωές ε, στη θάλασσα. Και αυτή είναι μια αναπόδραστη υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα διαρθρωτικά αίτια. Ε, και στη Μέση Ανατολή, στην Ιορδανία, στο Λίβανο. Έχουμε αυτή την ιδέα το σύμφωνο, του συμφώνου για να προχωρήσουμε και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και την Αφρικανική Ήπειρο. Και εγώ ως Πορτογάλος γνωρίζω καλά την κατάσταση στην Αφρική. Και οι ροές ανθρώπων από την Αφρική θα είναι σημαντικές τις επόμενες εβδομάδες, ε, τις επόμενους, ε, τα επόμενα έτη. Δεν πρόκειται για συγκυριακή χρήση, θα είναι διαρθρωτική αυτή η κρίση των μεγάλων μεταναστευτικών ροών και από την Αφρική, γι' αυτό και θα πρέπει να επέμβουμε κυρίως στην υποσαχάριο Αφρική. Είναι στο σωστό δρόμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προτάσεις της. Και πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει επίσης ε, να εξετάσουν κατά πόσο θα πρέπει να ανοίξουν στο θέμα των προσφύγων, αλλά και να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κρίση. Νομίζω ότι είναι πολύ να τα μαντάτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας συγχαίρω θερμά ε, για την ε, πρότασή σας και τους δύο αντιπροέδρους, γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση. Για δύο λεπτά η κυρία Φαζόν. Ευχαριστώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα για μια ε, εταιρική σχέση με αφρικανικές χώρες. Αυτό είναι ενισχυτικό. Η φτώχεια στην Αφρική δεν προέκυψε χτες. Ε, και εύχομαι απλά να μην είναι πάρα πολύ αργά, γιατί δεν υπάρχει αλληλεγγύη ούτε μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Και δεν κάνουν βεβαίως οι χώρες αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί στην Αφρική. Και πράγματι δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα η μεταναστευτική κρίση. Εγώ υποστηρίζω την παγκόσμια αυτή προσέγγιση, αλλά αναρωτιέμαι ποια είναι αυτά τα οποία αναφέρατε ως ε, προτερήματα αλλά και κυρώσεις για τις χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν. Χρειαζόμαστε περισσότερες ε, επενδύσεις αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε ε, μόνο το βάρος στις αφρικανικές χώρες και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να πάνε τα ευρωπαϊκά χρήματα στα λάθος χέρια. Πρέπει να είμαστε αυστηροί για το ποιος λαμβάνει τα χρήματά μας και να έχουμε και τίμιους ε, εταίρους και σημαντικό είναι επίσης να έχουμε νόμιμες διόδους όπως αναφέρατε. Η Βαλκανική δίωδος έκλεισε θα έπρεπε να υπάρχουν λιγότεροι θάνατοι στην ε, Μεσόγειο, αλλά ανοίγουν ε, άλλες ε, διαδρομές. Βλέπουμε λοιπόν πως έχω μάθει μάλιστα πως στην Ελλάδα είναι δυνατή η υποβολή της ασύλου μόνο μέσω Skype. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια στρατηγική προσέγγιση. Δεν είναι δυνατόν μόνο να σταματάμε τις ροές, πρέπει να υπάρχει και μια ειλικρινής συνεργασία με την Αφρική και να υπάρχει καλύτερη ανθρώπινη επαφή. Το δικαίωμα της μπλε κάρτας ο κύριος Φόικτ, από ό,τι με ενημερώνει οι συνεργάτες μου όμως εδώ κύριε Φόικτ, έχετε μιλήσει ήδη, επομένως θα σας επιφυλάξω την ίδια αντιμετώπιση που είχα και για τον κύριο Τελίτσκα. Έχουμε ήδη οκτώ μπλε κάρτες σε αυτή τη συζήτηση, καταλαβαίνω το ενδιαφέρον, αλλά έχουμε καθυστερήσει πολύ και έχουμε και πάρα πολλά αιτήματα για τη διαδικασία του Catch Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Κύρκος. Η εκρηκτική πληθυσμιακή ανάπτυξη της Αφρικής, σε συνδυασμό με την τεράστια φτώχεια ορισμένων περιοχών και με τους πολέμους, θέτει ένα καυτό ερώτημα. Μπορεί η μαζική, κατά εκατομμύρια μετανάστευση πολιτών από την Αφρική να αποτελέσει μέρος της λύσης. Η Επιτροπή με αφορμή την εισρωή δεκάδων χιλιάδων οικονομικών μεταναστών από την αφρική και όχι μόνο προσπαθεί να δώσει μια διπλή απάντηση και λέει όχι προτείνοντας ένα νέο φιλόδοξο πλαίσιο συνεργασία με κίνητρα και αντικίνητρα για τι χώρε τη Αφρική και τη γειτονιά μα. προσπαθεί να δώσει δηλαδή μια διπλή απάντηση και στην υπανάπτυξη αλλά και στη μείωση των μεταναστευτικών ροών. εάν μα πείσετε ότι με το σχέδιο αυτό θα χτυπηθεί η τεράστια κατασπατάληση πόρων και διαφθορά στην υλοποίηση των δράσεων μέσω ενός μηχανισμού διαφάνειας αλλά και ουσιαστικής διερεύνησης των καταγγελιών από την κοινωνία των πολιτών πιστεύω ότι η πρότασή σας θα αποτελέσει μια πολύτιμη συνεισφορά. αλλιώς κινδυνεύουμε να μιλάμε για ένα μηχανισμό συνδιαλλαγής με αξιωματούχους των αφρικανικών χωρών οι οποίοι θα αυξάνουν τα προνόμια τους ενώ η ευρώπη θα τους πληρώνει για να δέχονται τους πολίτες τους πίσω. ευχαριστώ. Ε, εγώ ευχαριστώ. Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών ολοκληρώνεται με την κυρία Σλάιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι χρειάζεται ένα σχέδιο επενδύσεων για την Αφρική μέσα στα πλαίσια της γενικότερης συνεργασίας. Φαίνεται όμως ότι στην ουσία ενισχύουμε τις τρίτες χώρες για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αποφύγουν τους πολέμους. Όμως η όλη έκθεση με τις τρίτες χώρες θα πρέπει να βασίζεται σε μία αμφίδρομη σχέση. Μιλάμε για επενδύσεις στην ουσία για διαχείριση των συνόρων, για border management, κάτι το οποίο αυξάνει τις ανισότητες και δεν αντιμετωπίζει τα αίτια των μεταναστευτικών ορών, γιατί και τις, τη βοήθεια που ζητήσαμε δεν την λάβαμε δεν έχει νόημα μόνο να υπερασπιστούμε τα εξωτερικά μας ε, σύνορα. Αυτό δεν αντιμετωπίζει τα αίτια του κακού. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών και προχωρούμε στην διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχτεί 17 αιτήματα με τη διαδικασία του Catch the Eye, όπως αντιλαμβάνεστε είναι αδύνατο να εικονοποιηθούν όλα. Θα δεχθώ τα πέντε από αυτά, ένα για κάθε πολιτική ομάδα, με βάση ως την σειρά καταγραφής όπως την κατέγραψαν οι συνεργάτες μου. Το λόγο έχει ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Άκουσα από την αρχή τη συζήτηση και την παρακολούθησα. Είναι πολύ επίμαχο και αφιλεγόμενο το θέμα και η συζήτηση το ίδιο ήταν αρκετά αμφισφόδρη. Πάντως ε, θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αν θέλει να αντιμετωπίσει αυτό το δύσκολο ε, θέμα και απαιτητικό θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο που μερικές φορές δεν ε, υπάρχει. Φυσικά έχει νόημα εταιρική σχέση με τι αφρικανικέ χώρε και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως μόχλευση την αναπτυξιακή και εμπορική πολιτική. Επίση, θα πρέπει να βάλουμε κάποια τάξη ε, στην κατάσταση, να ρυθμίσουμε την νόμιμη μετανάστευση και να καταπολεμήσουμε την παράτυπη. Επίσης να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι το θέμα αυτό είναι παγκόσμιο. Το πρόβλημα ε, δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και για το COP21 θέλουμε και για την μετανάστευση μια παγκόσμια λύση για να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα το θέμα και κυρίως να βοηθήσουμε εκείνους που προσπαθούν να γλιτώσουν από πόλεμο. Σα ευχαριστώ. Τρία χρόνια είμαι Ευρωβουλευτής και ακούω εδώ και τρία χρόνια για τη μετανάστευση και τα προβλήματα που δημιουργεί. Ε, δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μέλλον για τους ανθρώπους αυτούς στις χώρες τους ε, ε, και ούτε καταφέραμε να τους σώσουμε από θάνατο, από πνιγμό στη Μεσόγειο ούτε να αποφύγουμε τα προβλήματα εξαιτία τη ανεξέλεκτη παράτυπη μετανάστευση. Πάντως με ικανοποίηση άκουσα τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικεντρώνεται σε προγράμματα ενίσχυσης προ τι αφρικανικές χώρες και επενδύσεις. Είναι πολύ χρήσιμες οι επενδύσεις και η οικονομική βοήθεια. Αλλά προσοχή, αυτά τα δισεκατομμύρια επενδύσεις και τη βοήθεια θα πρέπει να φτάσουν σε εσφαλμένους δικαιούχους, να βοηθήσουν τους πολίτες. Αλλιώς θα είναι ανεπίλητο το πρόβλημα. Έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Κύριε εκπρόσωποι της Επιτροπής, οι προτάσεις της Επιτροπής θα μπορούσαν ε, να θεωρηθούν μεγάλη αποτυχία. Είπατε ότι μπορούμε να καλωσορίσουμε όλους τους μετανάστες γιατί είπαν ότι είναι πρόσφυγες, αλλά οι περισσότεροι είναι παράνομοι. Μιλήσατε για ε, μια κλίδα κατανομής που θα μπορούσαν να ήταν μόνιμη ή προσωρινή. Τίποτα όμως δεν έγινε. Μετά αποτύχατε με το δικτάτορα Ερτογάν κάνετε μια συμφωνία με έναν δικτάτορα ο οποίος κατατροπώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν τα σέβεται, δεν τα τηρεί. Επίσης υποσχεθήκατε να καταβάλλετε δισεκατομμύρια ως λίτρα σε αυτό το δικτάτορα, τον Ερντογάν. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που λένε που, ότι μπορούμε να καλωσορίσουμε όλους τους μετανάστες. Πάρτε το σπίτι σας τότε. Κυρία Ντεσσαρνέζ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Εδώ βρισκόμαι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ταυτόχρονα όμω μείναμε με την όρεξη. Γιατί θα πρέπει να έχουμε μια σαφή στρατηγική στην Ευρώπη και ένα σαφέ όραμα, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Έχουμε περισσότερο την αίσθηση ότι μάλλον υφιστάμεθα την κατάσταση παρά δρούμε. Θα πρέπει καταρχήν να έχουμε μια γνήσια σωστή πολιτική ανάπτυξης δεν χρειάζεται απλώ να λέμε ότι είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητέ στην Αφρική. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε την αναπτυξιακή μα πολιτική, γιατί να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί, κάτι που δεν ισχύει μέχρι τώρα. Δεύτερον, θα πρέπει να φτιάξουμε νόμιμε διόδου για την οικονομική μετανάστευση, νόμιμε οδού. Μόνο έτσι θα καταπολεμήσουμε την παράτυπη, παράνομη μετανάστευση. Θα πρέπει να δώσουμε ε, θεωρήσει ώστε να μπορεί να έρχεται ένα μετανάστη, να εργάζεται μερικού μήνε, να επιστρέφει και να επανέρχεται όταν υπάρχει απασχόληση. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε ε, εργοδότες που στην Γεωργία απασχολούν παράνομα παράτυπους μετανάστες. Επίσης να επιτρέψουμε ε, αποτελεσματική επανεισδοχή. Με τέτοιες αμφίδρομες ε, συμφωνίες θα μπορέσουμε ενδεχομένω να δώσουμε μια λύση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κυρία Μογκερίνη, κύριε Τίμερμας, ξέρω ότι έχετε καλή θέληση, αλλά η ρητορία δεν αρκεί. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για μια μειοπική στάση των κρατών μελών. Γνωρίζουν ότι οι πρόσφυγες πνίγονται στη θάλασσα και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Αφρική για την Αφρική. Το ξέρετε εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν κάνατε ε, τίποτα ή κάνατε υπερβολικά πολλά. Πώς θα επιτύχει η Επιτροπή τα κράτη-μέλη να αλλάξουν την εξωτερική, εμπορική και πολιτιστική τους πολιτική, καθώς και στρατιωτική έναντι της Αφρικής. Διαφορετικά δεν θα μπορεί να υπάρξει κανένας είδου συμμαχία. Ολοκληρώσαμε και τη διαδικασία του Catch the Τώρα το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής η Αντιπρόεδρος κυρία Μογκερίνη. Thank Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πολλές φορές ακούγοντας τα σχόλια θα ήθελα να είμαι ειλικρινής. Ίσως θα ήταν χρήσιμη μία σωστή ανάγνωση της πρότασης στη συζήτηση. Ε, σήμερα το απόγευμα έγινε μία πρόσμιξη πραγμάτων. Δεν πρόκειται για επικάλυψη της συμφωνίας με την Τουρκία. Τα δύο πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως είπε η Γαλλία στην αρχή, από την Τουρκία έχουμε Σύριους πρόσφυγες οι οποίοι ε, εργάζονται προσωρινά. Μιλάμε όμως για πρόσφυγες ε, που ετούνται άσυλο και αυτό εμπίπτει στο διεθνές ε, πλαίσιο αντιμετώπισης. Και θα χρησιμοποιήσω μία λέξη που δεν μου αρέσει. Αλλά έχουμε να κάνουμε με μία κατεπίγουσα ανάγκη. Τώρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Με την Αφρική έχουμε κοινά συμφέροντα και θα πρέπει να συνεργαστούμε για την ανάπτυξη της Υπήρου εταιρικά. Εσείς είπατε πώς ε, αντιδρούν οι συνομιλητές από την Αφρική. Μα πολύ καλά. Χτες ήμουν στη Νέα Υόρκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι αφρικανικές χώρες και οι χώρες από τη Λατινική Αμερική είπαν ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος, διότι δεν επενδύεται μόνο στην ανάπτυξη, κάτι το οποίο καταρχήν είναι σωστό και είμαι υπερήφανη γι' αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος δωρητής παγκοσμίω. και είμαστε και ο πρώτος δωρητής στην Αφρική και διεθνώς. Με το ίμιση της διεθνούς ε, ε, αρρωγής 68 δις και 20 δις κάθε χρόνο στην Αφρική. Είμαι υπερήφανη γι' αυτό και αυτό είναι ο σωστός δρόμος, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πηγαίνετε στην Αιθιοπία και συζητήστε με τις γυναίκες που επέστρεψαν από τον ε, Περσικό κόλπο όπου είχαν μετατραπεί σε σκλάβες και από το ΔΟΕ είπαμε ότι θα πρέπει να τους δώσουμε βοήθεια. Το συμφωνήσαμε με το ΔΟΕ. Τι κάνουμε. Στην ουσία προστατεύουμε τη ζωή τους, τις ζωές τους. Μιλήστε με τις ε, νέες γυναίκες από την Ιγυρία που ε, έγιναν ιερόδουλες στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τις ζωές τους, τη ζωή τους. Δεν προστατεύετε τους ανθρώπους όταν τους σώζετε από πνιγμό, αλλά και στην αρχή της ιστορίας τους. Πηγαίνετε στη Λαμπεντούζα να ακούσετε τι μας ε, λένε αυτές που επέζησαν. Δείτε το έργο Φόκο Αλμάρε, το οποίο παρουσιάστηκε και στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούστε τα λόγια τους. Λένε ότι έχουν μετατραπεί σε σκλάβους στην αρχή του ταξιδιού τους. Είναι αλυσοδεμένοι, βρίσκονται ε, κλειδωμένοι στις φυλακές και στα μπάρια των πλοίων. Έχουμε ανθρώπινη ευθύνη και αυτό αφορά και τους Αφρικανούς εταίρους. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη ζωή τους. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με διεθνείς οργανισμούς. Μέσα στα πλαίσια και της ε, είπα αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Μιλάμε για δημιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες. Πηγαίνετε στο Αγκαντές που ζούσε από τον τουρισμό πριν, γίνει, πριν καταστεί αυτό αδύνατον. Δώστε σε αυτούς τους νέους ευκαιρίες που δεν σχετίζονται με εγκληματικές οργανώσεις ή διακινητές. Ας εργαζόμαστε, ας εργαστούμε για την κοινωνική ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την προστασία αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Αρκεί αυτό, όχι φυσικά αλλά αν δεν αρχίσουμε να κάνουμε το σωστό, σε δέκα χρόνια αυτοί που θα έρθουν μετά από μας θα αντιμετωπίσουν τα ίδια. Και ελπίζω να είχαν προτείνει πριν δέκα χρόνια οι άνθρωποι που βρίσκονται στη δική μας θέση, αυτά προτείνουμε εμείς σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η πρόταση δεν θα αναστρέψει την κατάσταση σε 24 ώρες, αλλά καμία πολιτική δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Και θα, δεν θα πρέπει να πουλάμε όνειρα και αυταπάτες τους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν καλά ζητήματα και θέματα που μπορούμε να προωθήσουμε. Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Είναι μια καλή αρχή. Αυτό προτείνουμε λοιπόν σήμερα. Μιλάμε για άνοιγμα των σωστών διάβλων και διόδων για τη μετανάστευση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σύνεποι και φυσικά αυτό αφορά και άλλους διεθνείς φορείς και χώρες από την Ασία, από, το Ηνωμένο, από τα Ηνωμένα Έθνη, τη Λατινική Αμερική και την Αμερική. Δεν θα αλλάξουμε μόνο εμείς την Αφρική με το σύμφωνο αυτό, αλλά η αφρικανική ηγεσία θα το κάνει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αλλάξουμε τις αφρικανικές κοινωνίες. Βεβαίως θα γίνουν επενδύσεις, αλλά θα δημιουργηθούν και οι όροι για να μπορέσουν να καρποθούν σωστά αυτά τα μέτρα. Εάν θέλει κανείς να ε, κάνει μια πτήση από μια αφρικανική χώρα σε μια άλλη, πρέπει να το κάνει μέσω Ευρώπης. Με αυτό είναι λογικό. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν επενδύσεις, αλλά να δημιουργηθούν και οι όροι επένδυσης για να καρποθούν όλοι. Τη στιγμή που μειωθούν οι ροές στην ανατολική δίωδο ή οδό, βλέπουμε περισσότερες ροές στη Μεσόγειο. Μα πρόκειται για διαφορετικές ροές και διόδους. Μέσω της Λιβύης στη Σικελία πέρσι είχαμε πολλές ροές Σύριων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα. Δεν υπάρχει μετατόπιση, απλώς η Αφρική είναι μια νέα ήπειρος φτωχή, αντιμετωπίζει κλιματικές αλλαγές και είναι φυσικό να συμβεί κάτι τέτοιο αν δεν έχουμε μια μακροχρόνια στρατηγική και προοπτική. Αυτό σας προτείνουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει εξ ονόματος Επιτροπής επίσης ο Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, λίγες παρατηρήσεις μόνο έχω να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Μογκερίνη. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος πως ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε μια ανθρώπινη πολιτική προσφύγων είναι να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι χρήζουν διεθνούς προστασίας και ανθρώπων που έρχονται στην Ευρώπη γιατί βλέπουν ε, ότι εδώ υπάρχουν οικονομικές ευκαιρίες. Πολύ συχνά, και τα ακούσαμε και πάλι εδώ σήμερα, παριστάνουν οι άνθρωποι ότι όποιος φτάνει στις ακτές της Ευρώπης είναι οικονομικός μετανάστης. Άκουσα κάποιους που το είπαν σήμερα. Είναι ένας φτηνός τρόπος να ξεφορτωθεί κανείς τις ηθικές του ευθύνες απέναντι σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αλλά είναι δυνατόν όμως γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και όχι. Γιατί? Γιατί για πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα και η Ιταλία ε, αντιμετώπισαν το πρόβλημα μόνες και ζητούσαν ξανά και ξανά ευρωπαϊκές λύσεις και η μόνη απάντηση που λάμβαναν ήταν ότι δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι δικό σας πρόβλημα και κανονίστε το. Τώρα λοιπόν πρέπει να το λύσουμε. Και ο μόνος τρόπος να το λύσουμε είναι με έναν τρόπο ευρωπαϊκό και θα ε, μπορέσουμε να το λύσουμε και θα έχουμε πανευρωπαϊκή στήριξη για μια ανθρωπιστική πολιτική για τους πρόσφυγες εάν ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα της οικονομικής μετανάστευσης με τρόπο μειώσιμο. Και το σύμφωνο με τις αφρικανικές χώρες είναι ένα στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό πιστεύω πραγματικά πως ε, αυτή είναι η λύση. Δεν έχω ακούσει κανέναν από αυτούς που ασκούν κριτική να έχει καμιά καλύτερη ιδέα. Αν έχετε καμιά καλύτερη ιδέα, πείτε την. Το να λέτε να έρθουν όλοι είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να τελειώσει η ανθρωπιστική μας πολιτική. Να τελειώσει η υποδοχή προσφύγων στην Ευρώπη. Και ο πιο σύντομος τρόπος για να δώσουμε στους λαϊκιστές να πούν την ευκαιρία πως όλοι όσοι έρχονται εδώ πέρα είναι καιροσκόποι που ψάχνουν να μας εκμεταλλευτούν για ένα καλύτερο μέλλον. Πείτε το αυτό σε μια οικογένεια που φεύγει από τη Ράκα από το Χαλέπι. Πείτε τους ότι είναι οικονομική μετανάστες. Είναι σκάνδαλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι ως μέρος μιας τέτοιας μακροπρόθεσμης πολιτικής θα πρέπει να είναι το να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι θα επιστρέφουμε τους ανθρώπους στη χώρα προέλευσής τους εάν δεν έχουν δικαίωμα σε διεθνή προστασία. Και ακόμη σημαντικότερο, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες στις αφρικανικές χώρες για να μην εξαφανίζεται η βοήθειά μας στις τσέπες της ελίτ, αλλά να πηγαίνουν στους νέους που έχουν ταλέντο, να έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν τη ζωή τους στη χώρα τους. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και οπωσδήποτε δεν θα γίνουν αυτά από μόνα τους. Χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη και τη συνεισφορά τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ δεν είναι η έλλειψη χρηματοδότησης είναι ακριβώς το ότι δεν υπάρχει συντονισμός, ότι δεν κάνουν οι 28 τα ίδια πράγματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την ίδια κατεύθυνση. Αντί να έχουμε κάποιες ιδέες, ο καθένας τις δικές του επειδή είχε απικίες κτλ. Πρέπει να μπει μια τάξη. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανθρώπους. Δεν μιλάμε για νούμερα ή αντικείμενα. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν όνειρα, σαν και εμένα και εσάς, και θέλουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους. Που δεν θέλουν να τους εγκαταλείψει το πλούσιο κομμάτι του κόσμου. Και είχα μια εμπειρία την προηγούμενη εβδομάδα στη Σουηδία. Μια χώρα η οποία έχει δεχτεί κατά περισσότερους πρόσφυγες από οποιαδήποτε άλλη. Πάνω από 160.000. Τώρα έχουν, που έχουν την εντύπωση ότι σιγά σιγά το ελέγχουμε αλλάζει η διάθεση στην ε, Σουηδική κοινωνία και λένε εντάξει λοιπόν πρέπει να τα καταφέρουμε. Οι ε, εταιρείε προσφέρουν θέσεις μαθητείας, ε, τα σχολεία δέχονται μαθητές, οι κοινότητες καλωσορίζουν τους νέους πολίτες και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να δούμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Ζλάταν Ιμπραήμωβιτς ένα αστέρι γιος ανθρώπων που έφυγαν από την Βοσνία πριν από 25 χρόνια και είναι πολύ περήφανος που είναι Σουηδός και η Σουηδία είναι πολύ περήφανη γι' αυτό να δούμε πόσους Ζλάταν θα έχουμε σε 20 χρόνια Σουηδία Σας ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς και εσάς και την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Η συζήτηση έληξε. Επιτρέψτε μου πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα να σας